Καλημέρα σας. Καλημέρα σε αυτούς δηλαδή που έρχονται τώρα. Συνεχίζουμε με την ημερήσια διάταξη. Με το σημείο 16... Γιατί είναι για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις θαλάσσιες υποθέσεις και την αλία. Το Μάιο παρουσιάστηκε το έγγραφο εργασίας και θα προχωρήσουμε τώρα σε μια συζήτηση πιο σε βάθος για το περιεχόμενο και τους πολιτικούς προσανατολισμούς επί της ουσίας. Ο κύριος Καντέκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για τη δεύτερη ανταλλαγή απόψεων σχετικά ε, με το μελλοντικό αυτό ταμείο. Ε, βλέπω ότι ε, υπάρχουν αρκετοί βουλευτές οι οποίοι προφανώς έχουν φύγει ήδη διακοπές. Δεν πειράζει, θα συνεχίσουμε όσοι είμαστε. Ε, είχαμε ήδη μια πρώτη ανταλλαγή απόψε τον προηγούμενο μήνα στο έγγραφο εργασία μου ε, και τώρα ετοιμάζω και το σχέδιο γνωμοδότησης, το οποίο θα είναι έτοιμο σε λίγο. Έχει οριστεί την 24η Σεπτεμβρίου ε, η προθεσμία για τις τροπολογίες για να συζητηθεί τον Οκτώβρη. Όπως έχω πει επανειλημμένα, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι απαραδεκτή ως έχει και στρέφομαι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώ συγγνώμη, αλλά έτσι είναι, είναι απαράδεκτη. Επομένως, μέσω της εκθέσεως ε, θα, και μέσω των τροπολογιών επί του βασικού κανονισμού θα υπάρξουν ε, προθεσμίες, θα υπάρξουν αλλαγές. Όσον αφορά το μηχανισμό των ΜΑΠ, ε, έχουμε ε, πει ότι αναφέρονται στην ε, αγορά και εν πάση περιπτώσει ε, αυτοί που δεν έχουν διαβάσει καλά θα το θέμα θα ήθελα να τους παρακαλέσω, να τους ζητήσω να το πράξουν και να υπερψηφίσουν τις τροπολογίες μου για το τμήμα 4. Επίσης η διαφοροποίηση των αλληλευτικών δραστηριοτήτων είναι κάτι το οποίο κατά την άποψή μου είναι η ήπια και προγραμματισμένη ε, ε, και προγραμματισμένη απώλεια ή θάνατος καλύτερα της αλίας. Προχθές ε, είχαμε και μια ανταλλαγή απόψεων με την Κομισιόν και γι' αυτό στρέφουμε προς την Κομισιόν και τον ρωτώ. Πιστεύετε ότι πραγματικά οι αλίες θέλουν να καταλήψουν μια εργασία που θέλουν. Ξέρετε ότι ε, μονάχα 30% των προϊόντων αλληλείας και υδατοκαλλιέργειας που καταναλώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση παράγονται εδώ. Ε, και επίσης δεν έχω καταλάβει καλά τη λογική της εσωτερικής αγοράς. Ο προτινόμενος μηχανισμός είναι παράλογος κατά την άποψή μου οι παλιοί αλληλείς υποτίθεται ότι θα είναι ευνοούμενοι ε, σε σχέση με παλιούς ε, ε, φορείς της αγοράς. Ναι, αλλά τι γίνεται με τον σωστό ανταγωνισμό. Επίσης λέτε ότι θα πρέπει οι υδατοκαλλιέργειες να χρηματοδοτούνται από το Ταμείο. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν οι οι προϋποθέσεις για δημιουργία θέσεων απασχόληση κτλ. Επίσης, η Κομισιόν δεν αντιμετωπίζει τα πραγματικά προβλήματα της ε, ε, αλληλεία. α πούμε, γύρανση του αλληλευτικού στόλου. Τα περισσότερα πλοία είναι πάνω από 25 ε, ετών και επομένως τίθεται ένα ζήτημα προστασίας περιβάλλοντος και ασφάλειας. Προτείνω, πράγμα που έχω πει επανειλημμένα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο να βοηθήσει, να χρηματοδοτήσει τον εξυγχρονισμό ε, του ε, στόλου. Και επομένως ε, εγώ θα προτείνω να χρηματοδοτηθούν οι αγορές νέων πλοίων, νέων σκαφών, τα οποία θα είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον, θα είναι, πιο, θα είναι λιγότερο ενεργοβόρα κτλ. Χωρίς όμως ταυτόχρονη δυνατότητα αύξησης της ελληνική ικανότητας. Επίσης, ε, οι επαγγελματίες δεν ε, θα πρέπει να σταματούν τελείως ε, τις δραστηριότητές τους στη διάρκεια της βιολογικής παύσης ή στην διάρκεια των δυσμενών κλιματικών συνθήκων. Θα προτείνω λοιπόν, μία, θα προτείνω, λοιπόν κάποια μέτρα συνοδευτικά έτσι ώστε ε, να μην χάνουν εντελώ τον χρόνο τους ε, και ε, να μπορούν να συνεχίσουν κάποια δραστηριότητα οι αλληλείς κατά τη διάρκεια αυτών των παύσεων. Επίσης θα προτείνουμε κάποια εναλλακτικά μέτρα για την πάρα πολύ μεγάλη και απότομη αύξηση των, της τιμής των των καυσίμων. Στο άρθρο 41 επίσης θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές. Επίσης, εγώ θα προτείνω το άρθρο 41 να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του ε, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις Θαλάσσιες Υποθέσεις το άρθρο 70 ε, προβλέπεται ε, να είναι βαθμιαία ε, η διαγραφή μέχρι το 2016. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει το σύστημα αυτό. Θα πρέπει να βρεθεί ένα σύστημα το οποίο θα δώσει την δυνατότητα να δοθούν στην αγορά τα αποθέματα σε μια τιμή λογική και υποστηρικτική του εισοδήματος. Όσον αφορά την υδατοκαλλιέργεια, ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να παρέμβει το Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις Θαλάσσιες Υποθέσεις, όσον αφορά την βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια, ε, την σωστή επένδυση ε, για μια δραστηριότητα η οποία θα πρέπει να είναι συμπληρωματική και όχι ανταγωνιστική ως προς την θαλάσσια αλία. Ε, η ε, βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών οι οποίες ζουν από την αλία, ε, η χωροταξική ανάπτυξη και των, της ακτογραμμής και της, των θαλασσίων περιοχών είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, και βεβαίως ε, θα πρέπει ο τομέας της αλίας και της δατοκαλλιέργειας ε, να εκπροσωπείται σε όλες τις περιπτώσεις, έστω και αν σε μερικές περιπτώσεις όντως αυτό μπορεί να είναι περίπλοκο, συμφωνώ με την Επιτροπή. Όσον αφορά την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, 432 εκατομμύρια ευρώ προτείνονται αυτό σημαίνει τέσσερις φορές ε, ανά έτος ε, τον, ε, τον προϋπολογισμό που είχε μέχρι τώρα. Η χρηματοδότηση βεβαίως δεν θα πρέπει να γίνει προς ζημία της αρτοκαλλιέργειας και της αλίας. Γι' αυτό λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Ταμείο πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα όριο για το ΠΕΜΗ. Αυτά ήθελα να σας πω αγαπητοί συνάδελφοι. Το σημαντικό είναι ε, να δούμε ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο δεν θα είναι απλώς ένα εργαλείο μεταστροφής των αλλιέων όπως το βλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά ένα ταμείο το οποίο θα βοηθήσει την ανάπτυξη της αλλιείας, την σωστή ανάπτυξη. Ε, θα ήθελα το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις Θαλάσσιες Υποθέσεις και την Αλληλία να είναι λίγο εικονοκλαστικό. Δεν αμφιβάλλω καθόλου ότι ε, θα υπάρξουν παρατηρήσεις, ε, σχόλια και θα υποβάλλετε και τροπολογίες και βεβαίως εγώ θα είμαι πάντα στην διάθεσή σας να σας ακούσω αλλά και να συνεργαστώ μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Καντέκ. Το λόγο η Κομισιόν και μετά οι βουλευτές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να απαντήσω στα βασικά θέματα τα οποία έθεσε ο εισηγητής. Πρώτον, εγώ θέλω να καταστεί σαφές ότι για την Κομισιόν αυτός ο κανονισμός είναι ένας κανονισμός ο οποίος θα πρέπει να χρησιμοποιείται ουσιαστικά για να προωθήσει μία αλλαγή απαραίτητη για οποιαδήποτε πολιτική της αλίας. Ξέρετε ότι στο βασικό κανονισμό η Κομισιόν προτείνει ένα σωρό αλλαγές στην πολιτική. Εδώ προϋποτίθενται αλλαγές αλλιευτικών πρακτικών, ε, κλαδικές ε, προσπάθειες αλλά και κρατικές προσπάθειες. Και αυτός ο κανονισμός θέλει να δώσει την απαραίτητη υποστήριξη για να πραγματοποιήσουμε ουσιαστικά αυτές τις αλλαγές στην πολιτική που προτείνει η Κομισιόν. Άρθρο 32. Δεν θέλει να ε, να φορτσάρει τους αλλείς να εγκαταλείψουν την αλλιευτική τους δραστηριότητα, ούτε να παροπλήσουν πλοία. Αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει η Κομισιόν είναι να ορίσει στόχους μακροπρόθεσμα, αλλά δεν καταναγκάζει κανέναν να αλλάξει δουλειά. Θέλει να συνοδεύσει τον κλάδο και τις ε, κοινότητες που εξαρτώνται από την αλλιευτική δραστηριότητα. Και αυτό με την ιδέα ότι πρέπει να έχουμε μία ολοκληρωμένη ανάπτυξη, η οποία δεν αντιβαίνει με την αλία. Συμπληρωματική ανάπτυξη στην αλία. Όταν η Κομισιόν μιλάει για διαφοροποίηση, λέμε ότι πρέπει να προσθέσουμε στην αλληλευτική δραστηριότητα άλλες παράλληλες δραστηριότητες με εκείνες της αλίας. Εμείς δεν θέλουμε να εγκαταλείψουν το επάγγελμα του Αλία. Θέλουμε και άλλοι μέσα σε αυτές τις αλλιευτικές κοινότητες να ασκούν παράλληλες δραστηριότητες. Τώρα, για τη γύρανση του στόλου, ε, ναι, όντως υπάρχει πρόβλημα ηλικία των πλοίων. Γνωρίζουμε όμως ότι για τα τμήματα, για, για, τα τμήματα, για τους κλάδους εκείνους όπου έχουμε κέρδος από την αλία, ο στόλος ανανεώνεται τακτικά. Εκεί όπου έχουμε λοιπόν απόδοση στη, από την αλευτική δραστηριότητα, ανανεώνεται η, ε, ο, ο αλευτικός στόλος χωρίς να παρεμβαίνει το δημόσιο. Τώρα... Η εμπειρία που είχαμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι ο εξυγχρονισμός των πλοίων δεν σεβάστηκε πάντα την ιδέα της, του περιορισμού των ποσοτήτων αλληλευμάτων. Υπάρχει πρόβλημα στα κράτη με τον κυβισμό των μηχανών των πλοίων. και δεν μπορούμε εμείς να χρηματοδοτούμε τα πλοία για νέους κινητήρες όταν τα κράτη δεν έχουν υποέλεγχο την κινητήριο δύναμη. Και το πρόβλημα είναι βρει σε πολλές χώρες. Τώρα, για, τις για το εποχιακό σταμάτημα δραστηριοτήτων. Εμείς δεν προτείναμε αυτό το μέτρο, διότι έχουμε την τωρινή εμπειρία. Ξέρουμε ότι αυτά τα, αυτά τα κονδύλια υπάρχουν, αλλά η εμπειρία μας τόσο από την Κομισιόν όσο και από το ελεγκτικό συνέδριο μας λένε ότι τα κονδύλια ουσιαστικά δαπανώνται για να αντιμετωπιστούν κατεπήγοντα προβλήματα. αλλά κυρίως ε, για να τροφοδοτείτε με δημόσιο χρήμα στόλους οι οποίοι ούτως ή άλλως θα έπρεπε να διακόψουν στη συγκεκριμένη εποχή τη δραστηριότητά τους. Και αποτελεί δηλαδή μία επιπλέον πηγή εισοδήματος για τον κλάδο. Αυτός δεν είναι ο στόχος των διαρθρωτικών ταμείων, διότι τα διαρθρωτικά ταμεία λύνουν διαρθρωτικά προβλήματα, στην προκειμένη περίπτωση της και προτείναμε ακριβώς για να αξιοποιούνται σωστά τα κονδύλια να μην έχουμε κατά το επόμενο δημοσιονομικό έτος τέτοιου είδους κονδύλια. Τώρα, για τα λιμάνια. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι υποδομές των λιμανιών μπορεί να είναι ενδιαφέρουσες, αλλά ε, πολλές ε, λιμενικές ε, υποδομές σε ορισμένες ε, χώρες δεν λέω σε όλες, αλλά είναι μεγάλα. Εμείς έχουμε ένα σωρό γυροβόλια, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται σε πολλά λιμάνια. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς να συνεισφέρουμε σε μία σε μία υπερικανότητα Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε μία μεγαλύτερη ε, διείσδυση των διαρθρωτικών ταμείων. Ξέρουμε ότι ορισμένες υποδομές μπορούμε να τις χρηματοδοτούμε και με περιφερειακό ταμείο. Αλλά ε, αν έχουμε εμείς όμως περιορισμένα κονδύλια, τότε θα πρέπει να πασχίσουμε κονδύλια, ε, ε, υποδομές στην Αλία να πληρώνονται από το Περιφερειακό Ταμείο και να μην βγαίνουν χρήματα από, το, από, από την Αλία. Η ίδια λογική Ισχύει και για τη μεταποιητική βιομηχανία η οποία μπορεί να χρηματοδοτηθεί με άλλα κονδύλια και δεν χρειάζεται δηλαδή να ξοδεύουμε λεφτά της αλίας για την προκειμένη περίπτωση. Ε, εγώ το εξήγησα τώρα αλλά θα το ξαναπώ. Η βασική μας ιδέα είναι να δώσουμε ε, εξουσία αλλά και ε, ικανότητες ε, ε, στις ε, επαγγελματικέ οργανώσεις για να μπορούν να διαχειρίζονται την προσφορή. Και αυτό για να μπορέσουν οι οργανώσεις των αλλιέων να στήσουν μηχανισμούς και όταν αρχίσουν να λειτουργούν αυτοί οι μηχανισμοί να χρηματοδοτούνται από τις ίδιες τις ενώσεις συνεταιρισμούς των αλλιέων χωρίς να χρειάζονται δημόσιο χρήμα. Να χρηματοδοτούνται με ίδιους πόρους δηλαδή, για την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης. Σχετικά με την υδατοκαλλιέργεια, συμφωνώ με τον κύριο Καντέκ, που λέει ότι στόχος η, ναι, η υδατοκαλλιέργεια να είναι συμπληρωματική με την αλία. Δεν θέλουμε εμείς ε, να χρησιμοποιήσουμε την υδατοκαλλιέργεια ε, ως ε, εναλλακτική λύση γιατί δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τους σπόρους. Όχι. Συμπληρωματικά χρειάζεται δηλαδή καλή διαχείριση των αλλιευτικών πόρων και παράλληλα ανάπτυξη και της υδατοκαλλιέργειας. Διότι και οικονομική δραστηριότητα έχουμε κατά αυτόν τον τρόπο και πρωτεΐνες για τον κόσμο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε... Ευχαριστώ κύριε Πέρνας. Οχτώ ερωτήσεις έχω. Δύο λεπτά ο καθένας. Μάξιμουμ. Εννιά λοιπόν. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ απολύτως με αυτά που λέει ο κύριος Καντέκα ε, όσον αφορά την έκθεσή του, έστω και αν υπάρχουν κάποια σημεία επί των οποίων μπορούμε να βρούμε και κάποιες άλλες λύσεις. Πάντως, νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις Θαλάσσιες Υποθέσεις θα πρέπει να στηρίζει την πολιτική, κάποια πολιτική και όχι το αντίθετο. Ε, τα προτινόμενα των τον ΚΑΝΤΕΚ καταδεικνύουν συγκεκριμένο πρόβλημα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε το βασικό έγγραφο έτσι ώστε να έχουμε χρόνο για τις τροπολογίες ε, γιατί νομίζω ότι επανειλημμένα έχουμε από τους τελευταίους μήνες κάτι τέτοιο και θα ήθελα να σας καλέσω να σκεφτείτε στο ενδεχόμενο να ορίσουμε ε, προθεσμία για τις τροπολογίες μετά τις 24 Σεπτεμβρίου και μετά την ψηφοφορία του βασικού κανονισμού. Πιστεύω, ας πούμε, ότι όσον αφορά, το ευρωπαϊκό, όσον αφορά τις ε, ΜΑΠ, ε, θα ήθελα να καταλάβω αν υπάρχουν ναι ή όχι, γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν, η, η γνώμη του είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχουν. Αυτό σημαίνει ότι το συνολικό σύστημα που προτείνει η Επιτροπή που ε, βασίζεται στην ικανότητα μείω, μείωσης του ελευτικού στόλου βάσει αυτού του εικονικού μηχανισμού MAP, αλλάζει τελείως ε, την εικόνα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ποιο δρόμο ακολουθούμε. Πολύ σύντομα κιόλας, γιατί δύο λεπτά δεν είναι αρκετά για να πω όσα έχω να πω. Πιστεύω ότι θα πρέπει ε, να ε, δούμε το ενδεχόμενο του προγραμματισμού σαν ε, μια οδό την οποία ίσως θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε και βεβαίως ο πεπαλαιωμένος στόλος, ναι, όταν ένα στόλος έχει στην πλάτη του 35 χρόνια, προφανώς θα πρέπει κάτι να γίνει και θα πρέπει να υπάρξουν εξελίξεις, ας πούμε. Επίση, eh, Επίσης, ε, η, βιώσιμη, ε, συγγνώμη, η βιολογική παύση, ε, η οποία φαίνεται ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να δούμε όμως και ποιος είναι ο χώρος αυτής της παύσης. Λοιπόν, κύριε Μιλάνα, αλλά κυρία Φράγκα τώρα. Είναι άχρηστη όλη η συζήτηση. Όταν έχουμε εμείς ημερήσια διάταξη και 10-11 άνθρωποι ζητούν το λόγο, δεν μπορούμε να, χάσουμε το, να χάνουμε το χρόνο. 10 και 10 λοιπόν. 40 λεπτά. Είναι αδύνατον να τελειώνουμε την ημερήσια διάταξη. Κάλιστα να εντάξει, να, να καταργήσουμε σημεία. Να έχουμε περιορισμένα ημερήσιες διατάξεις. Να έχουμε πιο περιορισμένες ημερήσιες διατάξεις και περισσότερο χρόνο. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε εμείς τον κάθε ομιλητή 5-6 λεπτά ο καθένας. Λοιπόν, εγώ δέχομαι οποιαδήποτε πρότασή σας για το μέλλον, για το πώς θα οργανώσουμε τη δουλειά μας. Θα είναι πολύ καλές οι προτάσεις σας. Θα σας στείλω γράμμα, λέει ο κύριος Μιλάνα. Ευπρόσδεκτο, λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, εγώ θα ξαναπώ αυτό το οποίο είχαμε πει την πρώτη μέρα. Η απόσυρση των ενισχύσεων από τους τόλους έχει να κάνει με τον βασικό κανονισμό. Βασικός κανονισμός που πρέπει να είναι πιο αποδοτικός οικονομικά. Έχει δίκιο ο κύριος Πένα. Τώρα ε, επειδή το σχέδιο δεν ευόδωσε πουθενά ούτε στο Συμβούλιο ούτε στο Κοινοβούλιο κάτι πρέπει να βρούμε. Και εγώ λέω ότι δεν είμαι υπέρ των νέων ναυπηγήσεων πλοίων και αυτό που παρότι το εγκρίναμε χθες Φτάνει όμως να μην αλλάξει το μοντέλο διαχείρισης για τις ενισχύσεις αποθήκευσης. Εγώ συμφωνώ ότι μείωσε αρκετά τα μέσα παρέμβασης. Αλλά πρέπει να τελειώνουμε, διότι θα ήθελα μέχρι το 2020 να έχουμε την, την ενίσχυση για την αποθήκευση και αντί 1% της αξίας να είναι 2% της αξίας. Τώρα, ένα δις του ΦΕΠ θα πάει στην Κομισιόν σήμερα. Αλλά η Κομισιόν δεν παρουσιάζει τα ίδια προγράμματα εργασίας που παρουσιάζουν τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει λοιπόν η Κομισιόν να έχει τον αντίστοιχο σχεδιασμό με τα κράτη-μέλη. Τώρα για την υγιεινή και την ασφάλεια ενισχύσεις σε όλους τους αλλήλους και σε αυτούς ε, που ψαρεύουν με τράτες ε, και με, τις, σε, με όλες τις μεθόδους. Και συμφωνώ και με τον κύριο Καντέξ αυτό ότι πρέπει κάτι να κάνουμε. Τώρα για το 41 συμφωνώ υπέρ των αγκυροβολίων, διότι ορισμένες κοινότητες έχουν πολλά αγκυροβόλια ενώ άλλες λείπουνε. Το 86 Δεν θέλω να καταργήσουμε αυτό το 7% και πραγματικά εγώ με αυτές τις συνθήκες δεν μπορώ να δουλέψω. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ σημαντικό θέμα. Και μετά σε τρεις μέρες πρέπει να καταθέσουμε τροπολογίες. Ε, κύριε Πρόεδρε, πραγματικά δηλαδή. Ναι, αυτό για ορισμένους είναι το πιο σημαντικό θέμα της κοινοβουλευτικής θητείας. Για άλλους όχι. Είχαμε όμως ήδη συζήτηση. Είχαμε μια πρώτη συζήτηση. Δεν είχαμε ιδιαίτερο ενθουσιασμό από πολλούς. Αλλά αυτό το οποίο λέω είναι ότι η ημερήσια διάταξη αυτή που είναι. Και ο χρόνο είναι αυτό που είναι. Και αν θέλετε άλλη ημερήσια διάταξη, τότε να βγάλουμε δύο σημεία από την ημερήσια διάταξη σήμερα και άντε να συνεχίσουμε όσο θέλετε την κουβέντα. Αλλά εσεί δεν θα θελήσετε να βγάλουμε από την ημερήσια διάταξη. Ίσως μπορώ να προσφέρω εγώ μια ιδέα. Οι σκιώδεις ηγητέ θα έπρεπε να έχουν τουλάχιστον περισσότερο χρόνο από τους λοιπούς ομιλητές. Αυτό γίνεται και σε άλλες επιτροπές. Ίσως μπορούμε να δώσουμε ένα περιθώριο για μια τέτοια ιδέα. Α, υπολογίζεται αυτό στο χρόνο μου, ελπίζω όχι. Τώρα ξεκινάω λοιπόν τα σχόλια. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε πως θέλουμε μια άλλη Αλληλευτική πολιτική και πιστεύω ότι χρειάζεται πολύ χρήμα γι' αυτό. Πρέπει πολύ ευφυώς να αξιοποιηθεί το χρήμα που θα έχουμε και γι' αυτό πολλές από τις ε, προτάσεις του κυρίου Καντέκ μας βρίσκουν ε, σύμφωνους. Θα ήθελε παραδείγμα την επισημάνω ότι μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη χρειάζεται. Χρειάζεται η ε, κατάρτιση πάνω απ' όλα των εμπλεκομένων. Το είχαμε συζητήσει και στη Γαλλία και είχαμε επισημάνει ότι θέλουμε να δοθεί ευκαιρία στον Αλιέα που θέλει να εγκαταλείψει το επάγγελμα ή που οφείλει, που χρειάζεται να βρει μια διαφορετική λύση με διαφορετική κατάρτιση και επαναπροσδιορισμό ε, ε, των επιλογών του. Ξέρω ότι δεν έχω πολύ χρόνο για να συζητήσουμε διεξοδικά όλα τα προβλήματα. Είχαμε το θέμα των ε, διαλύσεων σκαφών, τα οποία δεν ήταν παλιά, δεν ήταν άχρηστα, ήταν καινούρια σκάφη, ήταν πιο ταχαία σκάφη και όμως ε, αναγκάστηκαν να προχωρήσουν στη διάλυση. Επίσης έχουμε να συζητήσουμε για ε, κανόνες όπου μπορούν τα κράτη να ε, ε, κάνουν κάποιες επιλογές για τη γεωργία με βάση το πρόγραμμα ε, ανάλογα με τις ανάγκες του αλλά να ε, υπαχθούμε στην, στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι υπερβολικό, μας περιορίζει υπερβολικά και δεν μπορούμε να έχουμε αρκετές δυνατότητες δεδομένων και των εξελίξεως στις τιμές των ορυκτών καυσίμων. Θα έχουμε αρκετά μέσα δηλαδή για να χρηματοδοτήσουμε τις δραστηριότητες. Επίσης θέλω να πω ότι εάν είναι καλά οργανωμένη μια δραστηριότητα και το έχουμε δει αυτό και στη Γερμανία και στη Γαλλία δεν χρειάζεται στήριξη και μπορεί η τιμή, οι τιμές του προϊόντος να διαμορφώνονται ανεξάρτητα ουδέτερα και χωρίς μειονεκτήματα. Η κρίση και η διαχείριση της κρίσης έρχεται ως ανάγκη όταν εμφανιστεί μόνο μια φυσική κρίση, μια φυσική καταστροφή δηλαδή και μόνο έτσι η καταβάση ή κατα... η επέμβαση ξέρουμε και το έχουμε δει στην Επιτροπή Γεωργίας ότι ουσιαστικά αυξάνει τις τιμές, δεν τις μειώνει. Κύριος Ρωμέβα. Και εγώ πάρα πολύ σύντομα. Είναι φανερό ότι όλα αυτά θα πρέπει να συνδέονται με το βασικό κανονισμό. Πρώτα πρέπει να έρθει το ένα και μετά το άλλο. Αλλά επειδή θα περάσει αυτό το στοιχείο της μεταφερόμενης ε, ποσόστοσης, θα πρέπει να συνδέσουμε το Ταμείο και με αυτό. Τώρα, υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Πρέπει να έχουμε μια διαχείριση αυτής της υπερικανότητας, ορισμένα μέτρα τα οποία δεν θα πρέπει να αντιβαίνουν σε αυτόν τον στόχο που είναι η μείωση της ε, ικανότητες. Δηλαδή δεν πρέπει εμείς να βελτιώνουμε την αλληλευτική μας ικανότητα αυξάνοντάς την. Αυτό είναι ένα από τα κεφάλαια που δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να τα τροποποιήσουμε. Τώρα αυτό που έλεγε η κυρία Ρόντους. Γι' αυτό εμείς επιμείναμε στο βασικό κανονισμό, στα κριτήρια. Κριτήρια δηλαδή για να είναι κανείς δικαιούχος. Αυτό που θεωρώ παράλογο είναι να ενισχύουμε την υπερκατανάλωση καυσίμων αντί να αμβλύνουμε τη δράση του, εκείνου του τμήματος του κλάδου το οποίο είναι ιδιαίτερα καψιμοβόρο. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να περιορίσουμε τα κίνητρα αυτών των δραστηριοτήτων. Τώρα, τα κεντρικά σημεία. Έλεγχος και επιστημονική ικανότητα, επιστημονική ανάλυση και επιστημονική έρευνα. Εγώ συμφωνώ να έχουμε αύξηση αυτής της ικανότητας, όχι μόνο για τον έλεγχο της κινητήριας δύναμης, που είναι ουσιαστικότατο, αλλά περισσότερο έλεγχο και στα λιμάνια και στην ανοιχτή θάλασσα και στον κλάδο. Και μία τελευταία αναφορά που ακόμη δεν βγήκε, αλλά συμφωνούμε με τον κύριο Μιλάν. Εγώ δεν θέλω να υποστηρίξουμε την υδατοκαλλιέργεια, αλλά θέλω να υποστηρίξουμε αυτούς τους προστατευμένους ηχθιότουπους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τον εισηγητή. Είναι προφανές ότι δεν συμμαριζόμαστε πολλές από τις ιδέες της έκθεσής σας. Πέραν των όσων είπε ο κύριος Ρωμέβα για τις ΜΑΠ δεν θα πρέπει να ενταχθούν πιστεύω στη χρηματοδότηση του ΜΦΕΦ αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι το ψάρι είναι κοινό πόρος, ανήκει σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και μόνο κακή διαχείριση των αλληλευτικών ε, αποθεμάτων έχει οδηγήσει σε μείωση των αποθεμάτων, σε κρίση σε κάθε κλάδο της ε, αλληλευτικής δραστηριότητας και λιγότερα ψάρια από τις ευρωπαϊκές θάλασσες στον ψαρά. Γι' αυτό λοιπόν αυτό που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι η υπερβολική αλλιευτική δραστηριότητα. Θα αντιμετωπίσουμε εάν την ελέγξουμε, εάν την περιορίσουμε και τα αποθέματα ε, και τις θάλασσες. Με τις ε, επιδοτήσεις δεν πρόκειται να βρούμε λύση, θα κάνουμε μάλλον κακό. Θα βρούμε μια βιώσιμη λύση για τον Αλιέα, γιατί θα έχει τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθεί και πάλι όταν αποκατασταθεί το αλληλευτικό απόθεμα και εξυγχρονιστεί ο στόλος. Πρέπει να δώσουμε δηλαδή τη δυνατότητα ακριβώς και τα χρήματα για την αποκατάσταση των αποθεμάτων και την παραμονή αλλιέων μέσα στο επάγγελμα μόνο κατά τρόπο ο οποίος να μην παραβλάπτει την ανασύσταση των αλληλευτικών αποθεμάτων. Για δε τις τιμές οι προτάσεις σας δεν είναι σωστές, δεν έχουν οδηγήσει σε λύσεις οι επεμβάσεις, οι παρεμβάσεις ποτέ στις τιμές, μόνο αυξάνουν την τιμή του προϊόντος, το οποίο αλλιεύεται κατά πλεονάζοντα τρόπο και στη συνέχεια πληρώνει ο Ευρωπαίος Φορολογούμενος μόνο και μόνο για να καταστρέφεται αυτό το πλεονάζον αλλιεύμα. και πιστεύω ότι όπως και η Ρόμπους θα οδηγηθούμε σε υψηλότερες τιμές μόνο. Επίσης θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν έχουμε να κάνουμε με αποτελεσματικότητα στη χρήση της ενέργειας των μηχανών των σκαφών, διότι και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πλεονόσολευτική δραστηριότητα. Ευχαριστώ, κυρία Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βεβαίως, όπως είπαν οι περισσότεροι και συμφωνώ, πρέπει να γίνει αυτό μέσα από την προσαρμογή της αλληλευτικής πολιτικής και από το βασικό κανονισμό βεβαίως το καταφέρουμε και θέλουμε να έχουμε ένα κλάδο αλληλευτικό ο οποίος θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, που θα έχει δηλαδή μια υπεύθυνη συμπεριφορά απέναντι στα αποθέματα, απέναντι στις αγορές, που θα πληρεί τις προϋποθέσεις και ταυτόχρονα θα ε, δίνει τη σταθερότητα που χρειάζεται τόσο στην απασχόληση όσο και στην οικονομική δραστηριότητα. Η πρόταση λοιπόν ε, της ε, πρόταση λοιπόν θα πρέπει να οδηγήσει την ανάπτυξη του κλάδου του αλληλευτικού κατά τρόπον βιώσιμο. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα για τα στοιχεία τα σχετικά με την καινοτομία που αναφέρει η έκθεσή σας Περιμένω να το, δω, να το βελτιώσω και εγώ με κάποιες τροπολογίες. Τη συλλογή επίσης δεδομένων. Θα ήθελα ακόμη περισσότερο να έχουμε κάποιες αναφορές στο πώς μπορεί να γίνεται η διαχείριση της, της θελάσσιας πολιτικής χωρίς να παρεμβαίνουμε στις αρμοδιότητες των κρατών, πράγμα το οποίο ξέρουμε ότι δεν έχει βοηθήσει ποτέ, το αποδεικνύει η ιστορία, ότι όποτε απλώς το μακρύ τη χέρι ε, το κέντρο, οι Βρυξέλλε δηλαδή δεν είχαμε καλά αποτελέσματα, αλλά πρέπει να γίνεται σε συνεργατικό μόνο τρόπο και όσο χρειάζεται. Επίσης, βλέπω ότι δεν υπάρχει επαρκής, επαρκώς ε, στέρεη ανάλυση αποτελέσματος και κόστους σε σχέση με τι προτάσει και εκεί χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια. Για δε το συνολικό προπολογισμό. Θα ήθελα να πω ότι ναι, μεν αντιλαμβάνομαι ότι έχει κάποιο νόημα να υποστηρίξουμε τιμέ κτλ. Έχει κάποια γοητεία ίσω το να κάνουμε τέτοιε προτάσει για επέμβαση. Αλλά δεν είναι αυτή η δουλειά μα. Η δουλειά μα είναι να δώσουμε τι προτεραιότητε ε, στην αλληλευτική πολιτική και τι προτεραιότητε δεν μπορούμε να τι δώσουμε κατά με σε ε, μια δραστηριότητα που είναι καθαρά ε, δαπάνη χρημάτων. Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε βοήθεια εκεί που χρειάζεται. Η κυρία Τόμα, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και δεδομένου του χρόνου που δεν έχουμε, θα ήθελα να επισέλθω στην ουσία των θεμάτων που με απασχολούν, ε, τα γενικά ζητήματα εν Συμφωνώ με τα περισσότερα από τα στοιχεία, τα σημεία που έχει αναπτύξει ο εισηγητής και ειδικότερα την ανάγκη να είμαστε προσεκτικοί ως προς το τμήμα αλληλεία και ενίσχυση της προτάσεις. Εγώ προτείνω να υποστηρίξουμε την, ε, το τμήμα της ολοκληρωμένης ελευτικής πολιτικής, όπως είπε και η κυρία Ρόντους, για την κατάρτιση αλλά και για την ε, εδαφική συνοχή, για τον προγραμματισμό τον, στο χώρο δηλαδή. Επίσης η έρευνα, η επιστημονική, η συλλογή δεδομένων πρέπει να λάβουν ιδιαίτερη προσοχή. Με στόχο βεβαίως την διαχείριση των αποθεμάτων έτσι ώστε να μην ε, πέσουμε στην ε, αυθαίρετη ουσιαστικά προσέγγιση της ε, αρχής της πρόληψης. Πρέπει να έχουμε στοιχεία ώστε να μπορούμε να ξέρουμε τι κάνουμε. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω ιδιαίτερα πόσο σημαντικός είναι ο έλεγχος στον προϋπολογισμό για να λειτουργεί σωστά το σύστημα. Για τα σκάφη συμφωνώ, όπως υπόθηκε και από την προλαλή σας, ότι θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στον εξυγχρονισμό, έμφαση στο βιώσιμο εξυγχρονισμό. Και όπως είπε και ο κύριος Πενιάς Λάντο, θα πρέπει να είναι διαρθρωτική η προσέγγιση αυτόν τον εξυγχρονισμό των σκαφών, διότι εάν θέλουμε επιλεκτικότητα για τα σκάφη, εάν θέλουμε πράγματι οικονομία και ως προς την προώθηση, και όχι σε ε, χρήματα μόνο, αλλά προώθηση ε, μηχανή, δηλαδή εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, ασφάλεια του ναυτικού, πάνω στο σκάφος, ε, γιατί ξέρουμε ότι γνωρίζει δυστυχώς αυτός ο τομέας πολλά, ακόμη και θανάσιμα ατυχήματα. Ε, εάν θέλουμε όλα αυτά λοιπόν πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι θα είναι αντιπαραγωγικό, ακόμη και αν ξέρουμε ότι θα πρέπει να επεξεργαστούμε το θέμα της υπερλεονάζως αλληλευτικής δυνατότητας. Θα ήταν αρνητικό για την αλληλεία να μην εξετάσουμε τη δυνατότητα να έχουμε στο μέλλον ένα σκάφος διαφορετικό, ένα καινούριο σκάφος, ένα σκάφος που θα πρέπει να χτίσουμε καινούριο για το μέλλον. Και για να χρησιμοποιήσω την ορολογία του κυρίου Πένιας Λάντος θα είναι πάρα πολύ δύσκολο αν θέλουμε να προχωρήσουμε στους ελέγχου στην ανιχνευσιμότητα, η χνηλασιμότητα, στην ε, διαχείριση της ε, μικρής κλίμακας ε, αλίας και εάν όλα αυτά, γιατί βέβαια δεν γνωρίζουμε θα είναι, ποιο θα είναι το μέλλον της μεταρρύθμισης, αλλά πάντως εάν η εκφόρτωση των ανεπιθύμητων αλλιευμάτων ε, έχει μια διαφορετική μεταχείριση. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε όλα αυτά. Έχουμε δηλαδή λειτουργούμενο κενό. Ευχαριστώ. Ελπίζω να μην μακρηγόρησα. Ο κύριος Γκρομπάσικ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω απολύτως με αυτά που είπε ο Όμως, ε, σε σχέση με την άποψη που εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πω το εξής. Μην λησμονούμε ότι υπάρχουν ε, κάποια στοιχεία περιοριστικά στον ε, κανονισμό. Ίσως ο καλύτερος τρόπος ε, θα ήταν να τα δώσουμε όλα στους Κινέζους έτσι ώστε να βγάλουν λεφτά γιατί αυτοί ξέρουν να βγάζουν λεφτά με οτιδήποτε. Επίσης μην ξεχνούμε ότι υπάρχει και η απελευθέρωση των εξωτερικών αγορών. Έχουμε δράσεις λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όσον αφορά τους δασμούς. Μην το ξεχνούμε και αυτό. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι δυνατόν, δεν είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε ανταγωνιστικά τις εξωτερικές ε, ε, αγορές. Στην ε, Βαλτική θάλασσα έχουμε, ας πούμε, ε, ε, έχουμε βιομηχανική αλία όσον αφορά ορισμένα είδη και καμία περιβαλλοντική αρχή δεν προστατεύεται εκεί. Επίσης το θέμα των ανεπιθύμητων αλλιευμάτων και των απορρίψεων είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε przede wszystkim bezpieczeństwo o e, Λοιπόν, όσον αφορά τώρα την ασφάλεια, ε, τα, οι μηχανές, η, ικανότητα των ε, μηχανών, η ισχύ τους ε, και κατά πόσον σχετίζεται με την αύξηση των αλλιευμάτων και, όσο, και πόσο σχετίζεται με την ελευτική ε, ικανότητα Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι να μπορεί ε, το αλίευμα να μεταφερθεί γρήγορα ε, στο σημείο εκφόρτωσης. Ε, αυτό, αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε το σκάφος να τριγυρνάει γύρω-γύρω έτσι ώστε να μπορέσει να πιάσει έτσι μια ικανή ποσότητα αλίευματος. Πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Ευχαριστώ πολύ. Αρσένης. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα συμφωνήσω ότι δεν έχουν την ίδια βαρύτητα όλα τα σημεία της σημερινής μας ε, ημερήσια διάταξη το, το Ταμείο για τι ε, θαλάσσιες υποθέσεις και την Αλία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και πρέπει να του δώσουμε χρόνο. Ε, το θέμα της αρεσιμότητας ε, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή τα χρήματα θα πρέπει να δοθούν εκεί όπου γίνονται σεβαστές ε, οι σεβαστές προϋποθέσεις και οι κανόνες. Επίσης, συμφωνώ με τους κανόνες προστασίας της βιοπικιλότητας. Επίσης, θα ήθελα να εισάγω τροπολογίες όσον αφορά την ε, ε, στήριξη των ε, περιοχών ανάπτυξης της Πανίδας και της θαλάσσιας Παρινδίδας έτσι ώστε να διατηρηθεί το επάγγελμα του Ελέα στην ε, στις θάλασσές μας. Ε, επίσης, όπως είπε και η κυρία Τομάς και άλλοι, χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα για, τον, ε, για τη συλλογή στοιχείων, καθώς επίσης και για την επιβολή των μέτρων. Και βεβαίως θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα της πλεονάζουσας ικανότητας. Ξέρουμε ότι στα ΜΑΠ υπάρχουν αρκετά προβλήματα και αν γίνουν, γίνει αποδεκτό αυτό το σχήμα θα είναι σε εθελοντική βάση και στην ουσία δεν προβλέπονται συγκεκριμένα μέτρα για για μείωση της ε, ε, αλλιευτικής ικανότητας. Και αν ε, δεν συνοδευτεί η πρώτη επιτροπή και από κάποια άλλα στοιχεία, δεν θα έχουμε κάνει καλά τη δουλειά μας. Επίσης, έχω σημαντικές επιφυλάξεις όσον αφορά τη χρηματοδότηση των, των λιμένων. Ανάγκη υπάρχει ε, έτσι ώστε να χρηματοδοτηθούν συγκεκριμένες δραστηριότητες ε, μέσω πιλωτικών προγραμμάτων ενδεχομένως ε, που θα μας δώσουν τις, τους σωστούς προσανατολισμούς τους οποίους θα πρέπει και τις σωστές πορείες που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Όσον αφορά την υδατοκαλλιέργεια πιστεύω ότι δεν έχουμε τις απαραίτητες ρήτρες αηφορίας και επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να στηρίξουμε την διατήρηση της ε, ναυτικής ε, πολιτιστικής κληρονομιάς ε, και βεβαίως και την δυνατότητα συντήρησης και διατήρησης των παλαιών ξυλίνων σκαφών. Ευχαριστώ πολύ, Τόρβαλτ. Thank Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο-τρεις σύντομες παρατηρήσεις μόνο. Θα πρέπει νομίζω να αναθεωρήσουμε την αρχή της σχετικής σταθερότητας, η οποία οδηγεί σε μια ουσιαστική αστάθεια, γιατί ο καθένας επιδιώκει το δικό του όφελος, ως προς τον εξυγχρονισμό του στόλου. Σε εποχές λιτότητας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, πιστεύω, να αξιοποιήσουμε καλύτερα την, ε, τα χρήματα που παίρνουμε από τον Ευρωπαίο ε, Φορολογούμενο το ανέφερε η κυρία Ρόντουστ ήδη, για τη διάλυση του Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, μια ειδική του έκθεση πέρυσι, επισήμανε μάλλον πρικτές εικόνες σε σχέση με την ε, δραστηριότητα της διάλυσης των σκαφών. Λέει θα πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους, δεν δούλεψε το σύστημα αυτό σωστά. Πρέπει να φτάσουμε στην ουσία του προβλήματος και να καταστήσουμε πάλι ενδιαφέρουσα, ε, συμφέρουσα δηλαδή οικονομικά την αλληλεία. μια ε, βραβευμένη με το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας που είχε, είχε εκδώσει ένα βιβλίο με τίτλο Tragedy of the Commons, τραγωδία των, των κοινών με κεφαλαίο. Ε, αυτή λοιπόν είχε πει ότι πρέπει πάντοτε να βρίσκονται διαφορετικές λύσεις. Κύριο Καντέκα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τα μέλη της Επιτροπής ε, που πήραν το λόγο ε, για ένα θέμα όπως είναι αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις Αλλαγές Υποθέσεις και την Αλία που είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το οποίο κύριε Πρόεδρε ε, θα έπρεπε να είχαμε προβλέψει λίγο περισσότερο χρόνο επομένως το Σεπτέμβριο θα πρέπει να βρούμε το χρόνο έτσι ώστε να συζητήσουμε ε, περαιτέρω θα έχουμε και τις τροπολογίες τότε και θα έχουμε και το σχέδιο γνωμοδότησης και επομένως μπορούμε να συζητήσουμε επί της ουσίας δεν θα απαντήσω στον καθένα ξεχωριστά, ούτε και συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την οποία είχα ανταλλαγή απόψεων χθε ακόμα για το θέμα αυτό. Συμφωνώ απολύτω με κάποιε προτάσει, ε, τι οποίε μπορεί και να εξελίξει περαιτέρω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπω επίση συμφωνώ και με μερικά από αυτά που ανέφεραν ε, οι συνάδελφοι. Παραμένω πεπισμένο ότι Συνολικά, εάν η Κομισιόν μπορούσε να προτείνει ένα πιο ισορροπημένο και λιγότερο ζωσπαστικό κείμενο, ε, δεν θα είχαμε τέτοιο μεγάλο πρόβλημα. Ε, δεν θα ε, καλούμεθα τώρα να τετραγωνίσουμε τον κύκλο, γιατί περίπου αυτό αντιμετωπίζουμε τώρα. Διότι το κείμενο της Κομισιόν εξ αρχής δεν είναι αρκετά ισορροπημένο. Πάντως, χαιρετίζω την εργασία που έκαναν οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά το θέμα αυτό, γιατί ξέρω πολύ καλά τη δουλειά που έχουν κάνει Έχοντα έχοντας ανταλλάξει επανειλημμένα απόψη μαζί τους. Ε, δεν θέλω να παρεξηγηθούμε. Δεν συμφωνώ με την αύξηση της ε, ικανότητας ε, του στόλου. Αντιθέτως, ο πρώτος στόχος μας είναι η διατήρηση του αλλιευτικού πόρου. Γιατί όπως λέω πάντα, εάν δεν υπάρχουν ψάρια, δεν θα υπάρχουν και ψαράδες. Ε, δεν θα πρέπει βεβαίως να με κάποιες προτάσεις, αλλά από την άλλη πλευρά δεν θα πρέπει ε, να τις ε, διατυπώσουμε με τρόπο που να μην είναι σαφές αυτό που θέλουμε να πούμε. Επομένως λοιπόν εγώ θα κάνω κάποια πρόταση βάσει και των όσων σχολιάσατε κι εσείς έτσι ώστε να κάνω μια ισορροπημένη πρόταση με την οποία θα συμφωνήσουν οι περισσότεροι αν και δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό και το καταλάβατε ήδη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Καδέκ. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα. Και εκμεταλλεύουμε την ευκαιρία σήμερα, γιατί έχουμε 17 βουλευτέ. Αφήστε δε και του 4 αντιπροέδρου, πράγμα το οποίο δεν συνηθίζεται ιδιαίτερα σε αυτήν την επιτροπή. Και είναι καλό να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία. Βέβαια, κανονικά 50 είμαστε όλοι και όλοι, τακτικοί και αναπληρωματικοί, οπότε πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Εγώ σήμερα άκουσα ότι θέλετε παραπάνω χρόνο, ότι είναι αδύνατο να δουλεύουμε χθε. Και χθε κάποιο μα είπε, μα γιατί φέρναμε αυτό το θέμα εδώ πέρα να το συζητήσουμε που ήδη το είχαμε συζητήσει, άρα δεν άξιζε καν τον κόπο να το ξανασυζητήσουμε σήμερα. Βλέπετε λοιπόν πώ έχουν τα πράγματα και πρέπει ο πρόεδρο να αποφασίζει. Αλλά εσεί ίσω να μην ξέρετε πώ λειτουργούν τα πράγματα. κάνουν μία πρόβλεψη οι υπηρεσίες της ε, γραμματείας για το κάθε ζήτημα και είναι μία αντικειμενική χρονική πρόβλεψη. Και ε, συζητήσαμε δύο, ε, δύο, δύο φορές τώρα και μία τρίτη θα συζητήσουμε το Σεπτέμβριο. Και είπανε μισή ώρα. Εδώ όμως συζητήσαμε μία ώρα και 27 λεπτά το θέμα. Και εγώ δεν μπορώ, δεν να ξέρω πόσο θα μοιραστεί ο, χρό, χρόνος. Σήμερα έχουμε 17 βουλευτές, για άλλο θέμα έρχονται 4. Και είναι δύσκολο πάντα να γίνεται η πρόβλεψη, εγώ προσπαθώ να είμαι ευέλικτος. Όντας όμως ότι η τελευταία μέρα της συνεδρίασης και πρέπει να τελειώνουμε στις 12.30 δεν έχουμε τέτοιες επιλεκτικές δυνατότητες. Εμείς ποτέ δεν είχαμε αυτό το πρόβλημα. Και δεν δίνουμε παραπάνω χρόνο στους ε, Σάντου, διότι οι σαντού έχουν τη δυνατότητα να συζητάνε άπειρα με τον εισηγητή. Και στην προκειμένη περίπτωση ποτέ δεν είχαμε το πρόβλημα να περιορίζουμε τόσο πολύ το χρόνο. Επόμενο σημείο. 19 στην ημερήσια διάταξη. Διατήρηση των αλλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλασσίων οργανισμών. Ο κύριος Γκάλαχερ είναι εισηγητής, ακούσαμε 31 Μαΐου τον κλάδο. Θα δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν για να μας παρουσιάσει το αντικείμενο αυτής της πρότασης. Η Κομισιόν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είχαμε... Όχι κύριε Γκάλαχερ, όχι. Όχι εσείς. Εγώ έδωσα καταρχήν στον εκπρόσωπο της Κομισιόν το λόγο για να μας παρουσιάσει την πρόταση και μετά ε, ως εισηγητής παίρνετε το λόγο εσείς. Adelante. Σας ευχαριστώ πολύ και καλημέρα σε όλους. Θα προσπαθήσω να δώσω μια σύντομη εισαγωγή, σύγκριση σε αυτήν τόσο τεχνικού χαρακτήρα πρόταση που έχετε ενώπιόν σας. Ξέρω ότι ένας από τους στόχους μεταρρύθμισης είναι στο μέλλον να έχουμε λιγότερο τεχνικά ζητήματα να αντιμετωπίσουμε εδώ στις Βρυξέλλες, αλλά εν πάση περιπτώσει πρόκειται για ένα κανονισμό, θα τον θυμάστε, τον έχετε ήδη συζητήσει. Και απορρέει από την εγκατάλειψη των κανονισμών, ε, από τους κανονισμούς μάλλον, μια σειρά τεχνικών μέτρων από τους κανονισμούς για τα τάκ και τις ποσοστώσεις. Πρόκειται λοιπόν για κανόνες οι οποίοι παρατάθηκαν ως προς την ισχύ τους ε, από, τις, από τον Ιανουάριο του 2010 στον Ιούνιο του 2012. Πέρσι εσείς αποφασίσατε να τους δώσετε άλλους 18 μήνες, βέβαια σας είστε μέσα από το Συμβούλιο, και έτσι ε, ισχύουν μέχρι το τέλος τρέχοντος έτους. Αρχικά είχαμε σκεφτεί και ελπίσει ότι θα είχαμε εντωμεταξύ προλάβει να ολοκληρώσουμε τη μεταρρύθμιση τη κοινή ελευθερικής πολιτικής μέχρι το τέλος του έτους. Αυτό όμως δεν φαίνεται πιθανό τώρα και έτσι άλλη επιλογή δεν έχουμε παρά να διατηρήσουμε αυτά τα τεχνικά μέτρα κατά βάση. Για άλλη μια φορά. Η ιδέα μας λοιπόν και πρόταση είναι ότι δεν μπορούμε πλέον αυτά τα μέτρα να τα ονομάζουμε ε, μεταβατικά εφόσον διαρκώς παρατηρούμε την ισχύ τους και έτσι προτείνουμε τη συγχώνευσή τους μέσα στον κανονισμό 850 του 98 ώστε να καταστούν τμήμα ενός συνόλου τεχνικών μέτρων χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα γενεά τεχνικών μέτρων μετά τη μεταρρύθμιση τη κοινή αλληλευτική πολιτική. Το θέμα είναι ότι προ το παρόν δεν έχουμε αρκετά στοιχεία στη θέση μα ώστε να καταθέσουμε προτάσει για το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, δεδομένου ότι βρίσκεται να εξελίξει η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση τη ε, ΚΑΛΠ και ότι πολλέ είναι οι μεταβλητέ ε, που μπορεί να επηρεάσουν τι εξελίξει πάνω απ' όλα ή ε, περιφερειοποίηση που, από την οποία θα εξαρταθεί η λειτουργία των τεχνικών μέτρων μας στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής και ταυτόχρονα η υποχρέωση για απόρριψη που έχουμε για συζήτηση αυτή την εποχή. Ε, αυτά είναι τα τεχνικά θέματα λοιπόν που έχουμε και θα ξεκινήσουμε από το δεύτερο εξάμεινο του 2012 με διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους ε, φορεί και παράγοντες, διαβουλεύσεις με τα κράτη-μέλη κτλ. για τη διατύπωση το εις νέας γενεάς τεχνικών μέτρων. Πολύ σύντομα λοιπόν, για να σας εξηγήσω τι περιλαμβάνει αυτή η πρόταση, όπως ε, εξήγησα και νωρίτερα, πρέπει να μείνουν ενισχύ τα μέτρα αυτά, γιατί μπορεί να, έχουν, ε, μπορεί να περιλαμβάνουν σημαντικούς για τη διαφύλαξη των αποθεμάτων κανόνους, έχουν, κανόνες. Έχουμε τρεις βασικές ομάδες για την βιωσιμότητα και διατήρηση των αποθεμάτων, όλα τα μέτρα του 2000, της Natura 2000 για τη δυτική ακτή της Ιρλανδίας, για τα ανοιχτά της δυτικής ακτής της Ισπανίας, την, ε, τις ανοιχτές ε, θάλασσες, τα μέτρα ε, για τις ε, θαλάσσιες στήνες ε, στην ε, Βόρεια Θάλασσα και άλλα που δεν θα, προ... θα σας εκθέσω αναλυτικά γιατί είναι πολυτεχνικά. Επίσης έχουμε μια άλλη ομάδα μέτρων που συνιστούν ουσιαστικά εφαρμογή μεταφορά των όσων συμφωνήθηκαν στον ΕΦΚ με την προστασία ιδιαιτέρως των ευάλωτων οικοσυστημάτων και μια τρίτη ομάδα κανόνες που αφορούν παρεκκλήσεις από τον κανονισμό 850 ε, του 98 κρίσιμου χαρακτήρα και που θα πρέπει να διαφυλαχτούν. Όταν τελευταία φορά συστήσαμε την πρόταση για την παράταση της ισχύω αυτών των μεταβατικών μέτρων και κάθε φορά που είδαμε από τη ΣΤΕΚΘ μια θετική επιστημονική ε, πραγματογνωμοσύνη ε, την ακολουθήσαμε. Ο συνάδελφος, εάν έχουμε το χρόνο, θα σας δώσει πολύ σύντομα κάποιες ε, προτάσεις και νομίζω ότι θα δείτε και στον πίνακα τι ουσιαστικά έχει γίνει. Ένα άλλο θέμα που κάναμε ήταν να απαλείψουμε μέτρα τα οποία είναι προφανώς πεπαλαιωμένα και ανεφαντικημένου και από τον κανονισμό 850-98 και ε, και από τον παλαιότερο κανονισμό των μεταβατικών τεχνικών μέτρων, δηλαδή ένα ξεκαθάρισμα ουσιαστικά, δεδομένου ότι δεν είχαν λόγο ύπαρξη πλέον αυτά τα μέτρα και θεωρούσαμε σκόπιμο να τα απαλείψουμε. Και αν μου δίνετε την ευχαίρεια, ο Ντομινίκ μπορεί να σας εξηγήσει εν συντομία τα κύρια στοιχεία της προτάσεώς μας, ε, που απορρέουν βέβαια και από τις προτάσεις ε, τόσο του Κοινοβουλίου όσο και του Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκαν αυτές πέρσι για την εφαρμογή των τεχνικών μέτρων. Ευχαριστώ πολύ, Ευνέστο. Σε σχέση με τα όσα έχουμε συμπεριλάβει στο άρθρο 19, παράγραφος 3 και 32α είναι μέτρα τα οποία ε, ήδη ε, συμφωνούν με τα όσα είχαμε προτείνει το 2009, αλλά υπάρχουν και αυτά τα οποία δεν έχουν ήδη ενσωματωθεί ε, στον ε, κανονισμό και οπωσδήποτε θα πρέπει να μπουν στο νομοθέτημα. 29 Δέλτα σχετίζεται με τις ε, περιορισμένες ε, περιοχές. Εδώ έχουμε ε, μια σειρά, μια σειρά ειδών τα οποία δεν μπορούν να ελιευθούν με εργαλεία κλπ και επίσης μπορούμε να δώσουμε και κάποιες επιπλέον πληροφορίες. Έχουμε περιλάβει εδώ και το θέμα της ασφάλειας των δικτυών. Ε, επίσης ένα ζήτημα το οποίο είχαν θέσει και το ε, Κοινοβούλιο και κάποια μέρη ε, και κάποια κράτη-μέλη και εδώ έχουμε βάλει συγκεκριμένους κανόνες κοινής ελευθερικής πολιτικής όσον αφορά την ενδιάμεση αξιολόγηση. 38 50-39 τα πελαγικά ήδη έχουμε προβλέψει ε, κάποια, συγκεκριμένα μέτρα τα οποία δεν είχαν αλλάξει από τη δεκαετία του 60 ε, και σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει λόγος να διατηρηθεί η, απαγόρευση. Ε, επόμενο σημείο το οποίο σχετίζεται με την περιοχή XA μικρότερα ε, πλοία με υποδύναμη λιγότερη από 12 κιλοβάτα και επίσης ε, ένα άλλο που πρέπει να σημειώσει κανείς είναι το εξή, στο σημείο 1 ε, των αρχικών μεταβατικών τεχνικών μέτρων και ξέρω ότι σας κουράζω αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε στην περιφέρεια 2α ένας αποκλεισμός δεν υπάρχει επιστημονικός, επιστημονικό υπόβαθρο για αυτόν τον αποκλεισμό και επομένως έρεται. Αυτά είναι τα ε, κύρια σημεία τροπολογίας τα οποία έχουμε υποβάλει. Κύριε Γάλαχερ, εσείς, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και θέλω να ευχαριστώ την Επιτροπή για την επισκόπηση που παρουσίασαν σήμερα για την ε, πολύ γενική εξέδωση Ε, για τη γενική παρουσίαση λοιπόν των προτάσεών τους, όπως είπε, έχουμε μια σειρά από ε, τεχνικά μέτρα από τα μέσα περίπου του 2011 και μιλάμε για μεταφορά ή παράταση ισχύω των ε, μέτρων αυτών. Ε, υπόθηκε βέβαια από την Επιτροπή ότι υπήρχε η ελπίδα για εξασφάλιση ε, μεταρρυθμίσης της αλληλευτικής πολιτικής της νέα αλληλευτική πολιτική στο τέλο του 2012, αλλά μάλλον έως το τέλο του 2013, γιατί δεν πιστεύω ότι υπήρξε ποτέ πραγματικά ελπίδα ότι μέχρι το τέλος του 2012 θα υπήρχε κοινή αλληλευτική πολιτική μεταρρυθμισμένη. Εν πάση είμαστε ρεαλιστές και αισιόδοξοι στα όσα κάνουμε εδώ και α μην έχουμε τεχνικά μέτρα τα οποία επηρεάζουν την διαβίωση τόσων πολλών και μικρής κλίμακας ε, αλλιέων. Εγώ ως εισηγητής θα μπορούσα να βρω τον εύκολο δρόμο να πω ότι παρατείνονται τα μέτρα όλα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και μέχρι το 2014 γιατί μετά θα έχουμε την κοινή ελευτική πολιτική. Όχι όμως, οι πολιτικοί δεν έχουν έρθει να κάνουν αυτή τη δουλειά, έχουν έρθει να κάνουν τη δουλειά αυτή ε, να κάνουν τη δουλειά τους όπως οφείλουν και όπως θεωρούν το καλύτερο ε, για όφελος όχι μόνο του ΑΛΕΑ αλλά πάνω από όλα της βιωσιμότητας των ελευτικών αποθεμάτων. Δεν μπορώ δηλαδή να αφήσω τα τεχνικά μέτρα να ισχύουν μέχρι ότου εξαλειφθούν όλα τα αποθέματα. Το Συμβούλιο, η Επιτροπή ή το Κοινοβούλιο δεν είναι δυνατόν να περιχαρακώνονται σε κάποιες ε, θέσεις και να μένουν Τι Πρέπει να κοιτάμε τι προχωρεί. Ο διάλογος, ε, ο τριμερής όπως λέγεται διάλογος, μπορεί να δώσει αποτελέσματα εάν ο κάθε ένας από τους συμμετέχοντες δείξει διάθεση να κάνει υποχωρήσεις και παραχωρήσεις προς τους άλλους. Άρα, τα τεχνικά μέτρα διατήρησης δεν μπορούν να συμπεριλαμβάνονται πλέον στον ετήσιο κανονισμό για τις αλληλευτικές ευκαιρίες που δημοσιεύονται κάθε χρόνο μετά, την, μετά το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Άρα πρέπει τα μέτρα αυτά να υιοθετούνται υπό τη διαδικασία της συναπόφασης μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου και έτσι ο κανονισμός 1288 του 2009 που παρατείνει τα μέτρα κατά 18 μήνες ε, και έτσι καλύπτει την περίοδο από τον Ιούνιο του 2011 και μέχρι, μέχρι τον Ιούνιο του 2011 και πέραν αυτού στη συνέχεια με τον κανονισμό 579 του 2011 δόθηκε μια άλλη παράταση για ακόμη 18 μήνες που εκπνέει τον Οκτώβριο τρέχοντος έτους. Η κατάσταση είναι αυτή και η Επιτροπή αντιλαμβάνεται βεβαίω καθής ότι δεν είναι δυνατόν να δώσει περαιτέρω παράταση μεταβατικών μέτρων για 18 μήνες. Και έτσι προτείνει τη μεταρρύθμιση του αρχικού, του βασικού κανονισμού δηλαδή, η οποία ε, ανάγεται στο 1998 και αυτή τη λύση έχει βρει. Προτείνει στη συνέχεια μια πιο ουσιαστική εις βάθος αναθεώρηση ως λύση, αντικατάσταση δηλαδή του εγγράφου του 98 μετά την υιοθέτηση της νέας κοινή αλληλευτικής πολιτικής, το νωρίτερο το 2014, ίσως και 15 όπως πιστεύω εγώ, γιατί δεν θα μπορέσουμε νωρίτερα να δούμε ένα ουδέτερο ανανεωμένο και πλήρες σύνολο μέτρων σε λειτουργία. Εγώ, ως μέλος της Επιτροπής λοιπόν, θεωρώ καθήκον μου να επιφέρω τον ρεαλισμό, να εισαγαγώ τον ρεαλισμό στις προτάσεις αυτές. Η πρόταση προς την, Ευρω... την Επιτροπή μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η εξή. Έχουμε να κάνουμε με 31 διαφορετικά μέτρα στον κανονισμό. 6 παραρτήματα, 29 άρθρα και 6 παραρτήματα, με ε, ίσως απλή διατύπωση, αλλά πάντως συνέπειες για πάρα πολλούς. Υποστηρίζω κάποιες από τις αλλαγές αυτές που αναθεωρούν ε, πεπαλαιωμένα ή απαρχαιωμένα μέτρα, όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά ταυτόχρονα πιστεύω ότι θα πρέπει να διατυπωθούν κάποιες στοχευμένες ε, τροπολογίες για να αντιμετωπιστούν προβλήματα και λήψη του κανονισμού του 1998. Ζητήματα δηλαδή τα οποία πλέον δεν έχουν λόγο ύπαρξης και που μπορεί να προξενήσουν προσθέσεις δυσκολίες στον ε, χώρο της αλίας. Πρόκειται για μέτρα τα οποία πολλές φορές αντιβαίνουν στην στο δικό μας ιδεώδες που είναι η ε, βιώσιμη διαχείριση των αποθεμάτων. παραδείγματι, στον ε, χώρο 6-8, στην περιφέρεια 6-8 για τον ε, γάδο, τα μέτρα για τα παραλιεύματα είναι εσφαλμένα. Και έτσι περνάω στις προτάσεις για την περιφέρεια 6α στην περιοχή της Σκοτίας και σε ένα βαθμό τα βορειοδυτικά της Ιρλανδίας με τον περιορισμό για την ε, ε, αλία του γάδου, του, της υπόγλωσσας ε, και άλλων αντίστοιχων ειδών, σημειώνοντας ότι είναι χαμηλά τα αποθέματα του γάδου και ίσως να μας πούν και ε, οι ειδικοί ότι δεν υπάρχει πια γάδος εδώ και καιρό στην περιοχή αυτή. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να γίνουν τροπολογίες και πρέπει οι τροπολογίες να ακολουθήσουν προτάσεις επιστημονικές για να στηριχθούν απαράδεκτη συνέπεια των μέτρων και της αποτυχίας τους στο χώρο, στην περιοχή 6α. Είναι και σας παρακαλώ να, να δείτε με το μυαλό, την εικόνα στο βόρειο Ατλαντικό σκαφών που φτάνουν μέχρι 80 μίλια μακριά, μικρά σκάφη, πολύ μικρά σκάφη, χωρίς ε, πραγματική ε, πραγματικό αντίκτυπο ως προς ε, την διατήρηση των αποθεμάτων που αναγκάζονται να φύγουν μακριά 80 μίλια για να, βρουν, ε, για να μπορέσουν να λεύσουν νόμιμα. Και εδώ δεν μιλάμε ούτε για τη Μεσόγειο, ούτε για τη Βαλτική, ούτε για καμία λίμνη. Μιλάμε για τον Ατλαντικό. Πρέπει λοιπόν αυτή την απόσταση να την περιορίσουμε. Επίσης πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να βρούμε μια κατάλληλη διατύπωση και να διαγράψουμε τελείως την πρόταση μια πρόταση στην οποία βρίσκω αποτρόπαια πρέπει να σας πω προς τις συνέπειές της. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν έχουμε μια μικρή περιοχή στο 6α, βορειοδυτικές ακτές, για την προστασία του νεογνού του γάδου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει λάβει απόφαση να κλείσει το χώρο αυτό. Οι Ιρλανδικές όμως αρχές, κατόπιν συστάσεως των ε, αρμοδίων εκπροσώπων του κλάδου, είπαν ότι, ότι πρέπει να κλείσει η περιοχή τελείω για μια συγκεκριμένη περίοδο τη αναπαραγωγή. Κλείνει όμω ουσιαστικά για του Ιρλανδού γιατί δεν έχει ληφθεί απόφαση από το ευρωπαϊκό επίπεδο και έτσι μόνο οι Ιρλανδοί δεν μπορούν να ψαρέψουν εκεί ενώ όλα τα άλλα σκάφη μπορούν. Αυτό λοιπόν πρέπει να γενικευθεί γιατί είναι ένα σφάλμα το ότι δεν ε, συμπεριελήφθη στον κανονισμό του 98. Μπορεί δηλαδή κάθε άλλο ευρωπαϊκό σκάφο να αλλιεύει στην περιοχή αυτή του 6α αλλά ε, και να ε, θέτει σε κίνδυνο τη διαχείριση ε, τη βιώσιμη διαχείριση των ελευτικών αποθυμάτων. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα σημείο που γίνεται λόγος για εκρηκτική αύξηση των αποθεμάτων του γάδου στην ε, περιοχή 6α. Εδώ είχαμε πρόσφατα μέτρα, έκτακτα μέτρα, με κατάργηση της ε, πρόβλεψης για, την, για το παρεμπίπτον αλλίωμα, για να απο, τραπεί δηλαδή ε, το παρεμπίπτον αλίευμα και έτσι να μην παραβλάπτεται το απόθεμα του γάδου. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να κάνουμε κάτι, διότι δεν βλέπω, τουλάχιστον από όσα λένε οι κοινωνικοί σύμβουλοι μας, ότι μέτρα έκτακτα δεν μπορούν να συνεχίσουν για πάνω από τι δύο περιόδου για τι οποίες έχουν εισαχθεί. Τουλάχιστον έτσι λένε οι νομικέ υπηρεσίε. Σε αυτό αναφέρθηκε η Επιτροπή ήδη. Είπε δηλαδή ότι στο μέλλον μπορεί σε περιφερειακή βάση, περιφερειακή βάση γνώμη, να γίνεται αυτή η αντιμετώπιση. Γιατί να μην το ξεκινήσουμε όμω από τώρα αυτό. Γιατί να μην γίνεται από τώρα αυτή η περιφερειακή αντιμετώπιση και οι χώρε εκείνε τα μέλη εκείνα τη Ένωση που έχουν ιδιαίτερη ιδιαίτερο συμφέρον θέλουν να προστατεύσουν τη δική του περιοχή, τι δικέ του θάλασσε να μην μπορούν να διαχειρίζονται περιφερειακά το πρόβλημα. Και έτσι φτάνω και στην ανάγκη κατεπηγόντως να προχωρήσουμε προς την περιφερειακή προσέγγιση. Γιατί αν περιμένουμε την ολοκλήρωση τη περιφερειοποίησης, τότε θα ε, φτάσουμε περίπου μέχρι το 2015. Θα είναι πολύ αργά δηλαδή. Γι' αυτό θα πρότεινα ε, να προχωρήσουμε και βέβαια να οριστεί και προθεσμία. Εγώ ετοιμάζω την έκθεσή μου κάπου μέσα στο καλοκαίρι και θα είμαι με τις τροπολογίες μου και θα είμαι στη διάθεση των συναδέλφων της Επιτροπής για οποιαδήποτε πρόταση. Πάντως, λαμβανομένου υπόψη ότι εάν δεν έχουμε κάτι μέχρι το, τα τέλη Σεπτεμβρίου θα καταρρεύσουν τα πάντα, το να πούμε ότι μπορούμε να επιλύσουμε μερικά προβλήματα δημιουργώντας κάποια άλλα δεν είναι απαραίτητα λύση. Ας είμαστε λοιπόν ρεαλιστές και προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τα πραγματικά προβλήματα με ρεαλιστικό τρόπο. Ταυτόχρονα όμως θα έλεγα ότι και εγώ θα θεωρούσα ότι δεν έχω επιτελέσει σωστά το έργο μου εάν έλεγα στην, Ευρωπαϊκή στην Επιτροπή μας ε, να αποδεχθούμε αυτομάτως ε, τις 29 ε, τροπολογίες που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσα από τις οποίες είναι σημαντικές, άλλες ίσως πλέον και λιγότερο σημαντικές και να δώσουμε την παράταση αυτόματα. Γι' αυτό λοιπόν σε πνεύμα συμβασμού, σε πνεύμα συνεργασίας θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν να είμαστε έτοιμοι για τα τέλη του χρόνου, αλλά όχι πάση θυσία. Ευχαριστώ κύριος Χάκτον. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Για τις επεξηγήσεις ευχαριστώ τον εισηγητή. Η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή αναφέρθηκε στα σημεία τα οποία προτείνει εγώ. Θα πω αυτά που δεν ε, προτείνω. Για το 6α ας πούμε, ε, και το ξέρει πολύ καλά ο κύριος Γκάλαχατ, ε, η κατάσταση είναι διαφορετική. Γνωρίζουμε όλοι κάθε μέλος εδώ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που λέει ότι είναι αποφασισμένη να λάβει υπόψη χρηστικές αποφάσεις Όλοι λοιπόν διατείνονται ότι είναι αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των απορρίψεων και όλοι, συμπεριλαμβανομένες και της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπή, ε, διατείνεται ότι θέλει ε, να έχει αποκεντρωμένη διαχείριση των αποφάσεων, αλλά αν δει κανεί αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν τα ακολουθήσει, θα αποτύχει όχι μονάχα ε, ε, για λόγους ε, τεχνικούς, αλλά είναι προφανές ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει η πρόταση της Επιτροπής. Γιατί, γιατί άμεσο αποτέλεσμα Έγκριση της πρότασης αυτής, έτσι όπως έχει διατυπωθεί από την Κομισιόνα, θα ήταν ε, στην ουσία μεγάλο ποσοστό απόρριψης του ε, γάδου. Ένα, αυτό θα ήταν άμεσο αποτέλεσμα. Αυτό έχει ήδη αναγνωριστεί δύο φορές μάλιστα και για δύο εξάμηνες περιόδους ε, και απεδείχθη ότι είναι ε, επίγον ε, θέμα και άλλωστε ε, ε, γι' αυτό έγινε στην ουσία και ο κανονισμός, για να βγει ο γάδος από την σύσταση του αλλιεύματο. Ε, και ε, είπαμε ότι θα, πρέπει, έπρεπε να είχαν υπάρξει και ανανεώσεις αυτής της αφαίρεσης για δύο εξάμηνα Και τι έγινε τελικά, τίποτα δεν έμεινε. Είπαμε όλοι ότι θέλουμε μείωση των απορρίψεων, το δηλώσαμε όλοι. Απ' την άλλη πλευρά παραμένει επίγουσα η κατάσταση και από ό,τι φαίνεται ε, είμαστε έτοιμοι για δύο ακόμα χρόνια ε, ίδιας κατάστασης όσον αφορά τις απορρίψεις. Αυτό το έχουν ε, κατανοήσει πλέον όλοι. Ε, και στις ε, προτάσεις ε, για μέγιστα επιτρεπόμενα αλλιεύματα και ποσοστώσεις έχει παραμείνει η σύσταση αλλιευμάτων και οι προτάσεις ακριβώς ίδιες. Έχουν δηλαδή αγνοήσει την επίγουσα κατάσταση. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Όσον αφορά τώρα το πρόβλημα που έθιξε ο κ. Χάλα χαρακτηριστικά με το ποιοι τελικά είναι αυτοί οι οποίοι ζημιώνουν. Μα, το θέμα είναι όταν ε, μια απόφαση φύγει, πλήττει μονάχα ένα πολύ μικρό μέρος ε, σκαφών και ένα πολύ μικρό μέρος αλλιέων, ε, τι γίνεται, ίσως γιατί νομικά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, μα αυτό είναι πολιτικά απαράδεκτο και είναι ανόητο τελικά να κάνουμε τέτοια πράγματα όταν ταυτοχρόνως λέμε ότι προτιθέμεθα να τροποποιήσουμε την κοινή ελληνική πολιτική. Δηλαδή ταυτόχρονα να ε, να ε, εξακολουθούμε να εφαρμόζουμε τις ίδιες αποφάσεις οι οποίες δημιουργούν τα ίδια προβλήματα εδώ και πάρα πολύ καιρό και τελικά να υφίστανται κυρώσεις και να ζημιώνονται οι ίδιοι εδώ και χρόνια. Νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε βάσει αυτών που είπαμε ότι θέλουμε να κάνουμε, αυτά που έχουμε ήδη διατυπώσει εδώ ε, όσον αφορά την μελλοντική διαχείριση των ε, αποθεμάτων ε, και να το κάνουμε τώρα και να μην περιμένουμε να έχουν περάσει άλλα δύο χρόνια μαζικής απόρριψης αλλιευμάτων. Ευχαριστώ κυρία Φράγα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να έχουμε παράταση του κανονισμού. Άσχετα αν η Επιτροπή μας είπε, ότι, είπε κάποτε ότι δεν ήθελε παρατάσεις. Τέλος πάντων. Ας είμαστε υπεύθυνοι και ας συνεχίσουμε. Το κεφάλαιο για τα μέτρα σχετικά με τα απόβλητα Αυτή η πρόταση όμως, αυτή, αυτός ο κανονισμός ε, βασίστηκε στο άρθρο 860 της ΝΕΑΒ. Λοιπόν, θέλω να ξέρω γιατί εδώ πάμε μέσω του 850 και όχι μέσω των ειδικών κανονισμών ε, που έχουμε ε, ε, ψηφίσει μέσα στα πλαίσια των διεθνών συμφωνιών με την ΝΕΑΒ. Εγώ θέλω σίγουρα να βγάλουμε ξεπερασμένα πράγματα. Αλλά αυτά δεν θα έπρεπε να τα δεις πάλι σε ένα πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης μας λέει στη ζώνη 5 η τροποποίηση του μεγέθους του χταποδιού. Όπως ε, επίσης ε, και ενός Ιαπωνέζικου ψαριού για, την, για τον κέντρο αν, Ατλαντικό. Και λέει ότι την κρίνουμε αυτό για βιολογικούς λόγους. Για, τους υπόλοιπους, όμως, για τις υπόλοιπες όμως αλλαγές δεν υπάρχουν βιολογικοί καταναγκασμοί. Λοιπόν, ό,τι είναι υποχρεωτικό σύμφωνη αλλά ό,τι γίνεται καθαρά από, από από, από θρησκευτικό φανατισμό, τότε τι να κάνουμε. Θα έπρεπε λοιπόν να έχουμε σχετικά με αυτά τα μέτρα πιο αντικειμενικά κριτήρια. Κανένας άλλος δεν θέλει το λόγο ή η Κομισιόν για να απαντήσει. Ωραία. Δεν θα πω πολλά. Όμως, σε σχέση με το 6α, ε, με την περιφέρεια 6α, ε, η Κομισιόν κατανοεί ότι για κάποιες ε, χώρες μέλη και όπως και για κάποιους βουλευτές δημιουργείται πρόβλημα. Όσον αφορά τώρα τα επίγοντα, τα επίγοντα μέτρα, τα είχαμε μέχρι τον Φεβρουάριο και μετά ε, πρέπει να πω ότι η πρόταση ήρθε μετά την ε, απόφαση για επιμήκυνση. Ε, κάποια από τα επίγοντα μέτρα μπορούν να εγκατασταθούν πιο μόνιμα εάν δεν υπάρξει άλλη ενδιάμεση αξιολόγηση. Ξέρετε, υπάρχουν κάποια προβλήματα χρονοδιαγράμματος και ενδεχομένως και χρονικές επικαλύψεις. Δεν νομίζω ότι η Κομισιόν αντιτίθεται στις τροπολογίες εάν το Κοινοβούλιο πιστεύει ότι πραγματικά πρέπει να υπάρξει κάποια τροποποίηση εδώ. Και όσον αφορά την σύσταση του αλλιεύματος, ε, όντως μπορούν να ε, αφαιρεθούν κάποια είδη. Το, για το 6α δεν ε, παρίσταται ανάγκη για περαιτέρω τροποποίηση. Δηλαδή ήδη έχουμε εδώ ε, συμπερίληψη των ε, μικρών ε, σκαφών και αναφορά συγκεκριμένων ειδών. Δεν έχουμε, δεν έχουμε πρόβλεψη για μικρές μηχανότρατες με ανυψωτικά μηχανήματα, με ανυψωτικά εργαλεία ε, τα οποία θα πρέπει να σταματήσουν. Ε, επίσης ε, δεν υπάρχει καμία επίπτωση όσον αφορά τα αποθέματα των προστατευομένων ειδών και κάποιες εξαιρέσεις μπορεί να τις λάβει υπόψη της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά το χταπόδι και τα οστρακοειδή, χτένια κλπ. Ε, κάποια από τα μέτρα αυτά ε, απλώς έχουν, μετατε, με, έχουν αντιγραφτεί κατά κάποιο τρόπο από τα μεταβατικά ε, μέτρα. Είχαν ήδη προβληθεί το 2009, αλλά δεν είχαν ενσωματωθεί ποτέ σε νομοθεσία. Σχετικά με το κατά πόσον ε, οι βουλευτές θα ήθελαν ε, περαιτέρω εξηγήσει ε, για τα προβλεπόμενα εδώ. Βεβαίως μπορούμε να υποβάλλουμε περαιτέρω επεξηγήσεις και αρκετά γρήγορα. Ευχαριστώ. Εγώ αναρωτιέμαι. Είναι νορμάλ κατά τη γνώμη σας να μεταφέρετε αποφάσεις περιφερειακών οργανισμών στους, ε, στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία λέτε γιατί είναι κατεπήγον. Ωραία, αλλά δεν υπάρχουν οι δικοί μας ε, κανονισμοί που μας προστατεύουν. Εγώ θέλω να σιγουρευτώ, δεν καταλαβαίνω με τη διαδικασία, θέλω να σιγουρευτώ ότι αυτός είναι και ο μόνος λόγος δηλαδή που ενσωματώνουν αυτή την πρόταση. Κομισιόν απάντηση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία άλλη ειδικότερη απάντηση. Έτσι τα έχουμε κάνει. Δεν, ε, ε, ε, ξέρω τι άλλο να σας πω, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ήταν σαφές. λόγω κατεπήγοντος ή για άλλους λόγους. Ο κύριος Γκάλαχερ για να ολοκληρώνει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, για την ε, συμβολή της συζήτηση, ιδιαίτερα την ε, Κάρμεν Φράγο. Δεν μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις. Και δεν νομίζω ότι είμαι εγώ ικανότερος να δώσω απαντήσει από τη δική της Επιτροπής. Αλλά κάτι στο οποίο μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση είναι ότι έχουμε την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε το χρονικό ζήτημα μετά το 2009 και χαίρομαι για την ε, θέση της Επιτροπής που φαίνεται να λαμβάνει υπόψη την κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε. Και πιστεύω ειλικρινά ότι θέλουν να αξιολογήσουν την κατάσταση και ε, να τη δουν στις πραγματικές τους διαστάσεις. Επίσης, είμαι βέβαιος ότι θα αποδεχθούν το το Κοινοβούλιο δεν θα κάνει πρόταση για απλή παράταση της διάρκειας των ε, μέτρων. Κάποια έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μας, πρέπει να σας πω, για την ε, περιοχή 6α, ε, η οποία έχει μεγάλη σημασία για μας. Σκοτία και τα λοιπά, αλλά όχι μόνο αυτήν όχι μόνο αυτήν, είναι πολλά τα σημεία στο οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε μια υπεύθυνη στάση. Και αυτό που θα προτείνω δεν θα έχει λόγους μόνο δεν θα έχει λόγους πολιτικούς, δεν θα είναι πάνω σε βάση πολιτική, αλλά σε επιστημονική βάση, γιατί στην επιστημονική βάση στηριχθούμε για τις τροπολογίες μας. Ξέρω ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν είχε προβλεφθεί τα μέτρα, τα, τεχνικά αυτά μέτρα το Φεβρουάριο να μην μπορούν περαιτέρω να παραταθούν. Ξέρω ότι είναι η κατάσταση πολύ δύσκολη. Και αυτό προκύπτει μετά την κατάθεση των προτάσεων. Επίσης, σημειώνω με ικανοποίηση την παρατήρηση ότι δεν σκοπεύει η Επιτροπή να αναθεωρήσει το θέμα περί απάλληψης του ανταγωνισμού. Ελπίζω λοιπόν ε, να κατανοήσει η Επιτροπή ότι δεν μπορούμε ε, να προσπαθήσουμε να τα συμπεριλάβουμε όλα αυτά μέσα σε μια έκθεση, ότι δεν είναι δυνατόν να δεχθούμε αναφετέρου τις προτάσεις. Ξέρουμε ότι πρέπει μέχρι το τέλος του χρόνου να είμαστε έτοιμοι και σας διαβεβαιώ ότι θα έχω την έκθεσή μου έτοιμη με τις προτάσεις ώστε να γνωρίσει και η Επιτροπή ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα μας επακριβώς. Προτείνω λοιπόν, εάν Πρόεδρε συμφωνείτε και εσείς, στις 19 Σεπτεμβρίου να κάνω την παρουσίασή μου. Θα έχουμε μικρή προθεσμία μέχρι το από τότε για, προ, για τροπολογίες, για να προλάβουμε να ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας τον Οκτώβριο, στη συνεδρία του Οκτωβρίου της Επιτροπής και να πάμε στην τον Νοέμβριο, στη δεύτερη Ολομέλεια του Νοεμβρίου Εάν όμω δεν το προλάβουμε αυτό, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Και επαναλαμβάνω ότι μπορεί να επιληθούν κάποια προβλήματα, αλλά μην ξεχνάμε ότι αν επιληθούν κάποια προβλήματα, μπορεί ταυτόχρονα να δημιουργηθούν άλλα και περισσότερα. Και όλα αυτά θα τα έχουμε υπόψη, ετοιμάζοντα το κείμενο. Φαντάζομαι όμω ότι και η Επιτροπή θα πρέπει να τα λάβει αυτά υπόψη. Το γεγονό ότι υπάρχει ο κίνδυνος να ε, μην έχουμε λύσει μέχρι το τέλο του χρόνου, μας υποχρεώνει να εργαστούμε όσο το δυνατόν σκληρότερα και σε συνεργασία για να εξασφαλίσουμε μια λύση μέχρι το τέλος. Ευχαριστώ κύριε Γκάλαχερ. Έχει αποκατασταθεί η ηρεμία. Έχουμε μείνει λίγοι στην αίθουσα και ο πρόεδρος έχει μείνει μόνος του, χωρίς αντιπρόεδρου Βλέπετε πώς έχουν τα πράγματα. Πάμε τώρα στα θέματα ασφαλείας ε, των πλιαρίων που πρέπει να τους ε, βγάλουμε τα πτερή καρχαρία από δίπλα, ε, από τα πλευρά. Η κυρία Πατράου έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι λυπούμε πολύ για το αργοπορημένο τρόπο με τον οποίο ε, ε, αρχίσαμε να συζητούμε για το θέμα αυτό, για διάφορους λόγους βεβαίως, ε, ήταν άτυχη αυτή η έκθεση και στην πρώτη και στη δεύτερη ανταλλαγή απόψεων ε, στην ουσία ε, δεν είχαμε πια βουλευτές, ε, ήταν απόντες οι σκιώδες εισηγητές και τα λοιπά. Και τώρα είχε προβλεφθεί για χθες αυτή η συζήτηση, την αναβάλαμε για σήμερα, πάλι είμαστε λίγοι. Τι να πω. Εγώ έπρεπε να πάω στην Αυστρία και στην ε, ε, Ιταλία με την Επιτροπή Γεωργίας και αναγκάστηκα ε, να μείνω εδώ μόνο και μόνο για να παρουσιάσω την έκθεση αυτή. Εν πάση περιπτώσει, προσπάθησα να ε, δραχθώ της ευκαιρίας έτσι ώστε να κάνω και έτσι κάποια ε, ενδιαφέρουσα δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα. Ε, θα θυμάστε ενδεχομένως και το σεμινάριο του το, που οργανώσαμε πριν μερικού μήνες και εκεί είχαμε μεγάλη συμμετοχή και από τους κοιόδης εισηγητές Εν πάση περιπτώσει, ήταν ένα σεμινάριο το οποίο απεδείχθη ιδιαίτερα ενδιαφέρον και με τους ε, εκπροσώπους της Κομισιόν και με τους εκπροσώπους της Shark Alliance ε, και με τους ε, ενδιαφερόμενους και τους εργαζόμενους στον τομέα. Απεσαφηνίστη ότι η η αφαίρεση των πτερυγίων είναι μια συνήθις πρακτική κυρίως ε, στους μη ε, ευρωπαϊκούς στόλους ε, και βεβαίως η οικονομική και κοινωνική ζημία μπορεί να είναι μεγάλη και θα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας αν δώσουμε στήριξη και συνέχεια στην πρώτη της αναφέρομαι και σε οικονομικές ε, ζημίες και βεβαίως τις ταυτίζω ή μάλλον τις, ε, ε, αναφέρω μαζί με τις κοινωνικές ζημίες γιατί ξέρετε ότι αυτά πηγαίνουν μαζί. Από την άλλη πλευρά βεβαίως υπάρχουν και περιβαλλοντικές ζημίες. Εμείς περιμένουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία θα διασφαλίσει ότι ε, δεν ε, υπάρχει πλέον υποψία αφαίρεσης ε, πτερυγίων. Στο σεμινάριο κατέστησα σαφές από διάφορες παρεμβάσεις ότι εάν δεν συνεργαστούμε με τους εμπλεκόμενους δεν θα μπορέσουμε να έχουμε όλα τα στοιχεία τα οποία, και τα δεδομένα τα οποία μας χρειάζονται. Αυτό είναι κάτι ενδιαφέρον. Ε, κάτι άλλο το οποίο ε, είναι καλό να υπογραμμίσουμε είναι το εξής. Ε, αναφέρθηκε και σαφώς ότι οι ίδιοι οι πλειοκτήτες προτίθενται, είναι μάλλον, έχουν τη διάθεση να χρηματοδοτήσουν έναν οργανισμό ο οποίος ε, θα είναι υπεύθυνος ε, για τις εκφορτώσεις ε, στα λιμάνια. Λοιπόν, μεγάλη αργοπορία είπαμε στην παρουσίαση της έκθεσης που όμως μας έδωσε και την δυνατότητα, την ευκαιρία να ζητήσουμε ακόμα μία αξιολόγηση επιπτώσεων, μίας από μια μονάδα αξιολόγησης. Δεν ήξερα ότι υπήρχε αυτή. Η μια μονάδα λοιπόν που δημιουργήθηκε στο Κοινοβούλιο και που ασχολείται ε, με τις μελέτες αντικτύπου. Είναι μια ε, μονάδα η οποία παίρνοντας τις μελέτες αντικτύπου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει μια δική της αξιολόγηση. Εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτή η μονάδα στο Κοινοβούλιο τη στιγμή του σεμιναρίου, όμως είχα την πληροφόρηση αυτή εκ των υστέρων και επομένως ζήτησα μια γρήγορη ε, αξιολόγηση από την εν λόγω μονάδα. Ε, γιατί στην ουσία αυτοί ήθελαν ε, πολλούς μήνες ε, προθεσμία έτσι ώστε να κάνουν μια πραγματική και σε βάθος ανάλυση. Εγώ ζήτησα μια πρώτη ας πούμε εκτίμηση, μια πρώτη αξιολόγηση της, της εκτίμησης αντικτύπου της Επιτροπής έτσι ώστε να έχουμε μια ιδέα. Κάποια στοιχεία λοιπόν τα οποία ε, προκύπτουν από αυτήν την αρχική ε, αξιολόγηση, τη αξιολόγησης αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, μου φαίνονται πολύ ενδιαφέροντα. Υπάρχει μια πρώτη φράση, που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχεται ότι η ευρωπαϊκή στολή φαίνεται ότι έχουν λίγες απορρίψεις πτερυγίων. Καρχαρία. Και επομένως ο αντίκτυπος ε, στην ε, ε, διατήρηση αυτού του ελληνικού πόρου φαίνεται ότι είναι μικρή. Αυτό προκύπτει από την αξιολόγηση επιτροπής βεβαίως. Έτσι. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ε, ε, στη βάση της ε, πρώτης της Επιτροπής υπάρχει μία δημόσια κίνηση στην οποία ενδεχομένως δεν έχουν ληφθεί οι υπόψη όλα τα στοιχεία. Επίσης, το Συμβούλιο Αξιολόγησης επέκρινε τον, ε, τη μελέτη αντικτύπου γιατί δεν είχε λάβει υπόψη της όλα τα στοιχεία ε, ας πούμε όσον αφορά τις ελλειπείς ε, επιθεωρήσεις πρέπει επομένως ο έλεγχος να είναι πιο διαρκής και πιο αυστηρός ε, έτσι ώστε να αρθούν οι υποψίες για αφαίρεση πτερυγίων επί των σκαφών. Επομένως, ενίσχυση των επιθεωρήσεων. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κάνει ποσοτικό, ε, ποσοτική μελέτη του οικονομικού αντικτύπου ή μάλλον να διορθώσω του ε, οικονομικοκοινωνικού ε, αντικτύπου. Πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες αξιολογήσεις. Δεν μπορούμε εμείς να εγκρίνουμε νέα μέτρα χωρίς να γνωρίζουμε ε, ε, τα, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα τα οποία προκύπτουν. Ένα άλλο ζήτημα ε, βάσει της αξιολόγηση που έκανε η νέα μονάδα του Κοινοβουλίου αναφέρεται στην ορθή ανάλυση κόστους ωφέλους. Σύμφωνα λοιπόν με την μονάδα αυτή του Κοινοβουλίου δεν έχει υπάρξει σωστή μελέτη κόστους κόστους-οφέλους Επομένως, ε, ε, μια ποιοτική ανάλυση κόστους κόστους-οφέλους ε, τώρα λαμβάνει η χώρα και θα πρέπει βεβαίως να προχωρήσει έτσι ώστε να έχουμε όχι μόνο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά στοιχεία. Επίσης, όσον αφορά κάποια νέα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν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 της διαρκούς αναβολής ε, ε, της ε, εκθέσεως στην ουσία δυσκολευόμαστε να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα. Ακούστε, εγώ από την αρχή είχα πει ότι δεν μπορούμε να... Εμείς δεν έχουμε βούληση, ούτε διάθεση, ούτε πρόθεση να πάρουμε τη μία ή την άλλη πλευρά, να συμφωνήσουμε με τη μία ή την άλλη πλευρά. Εμείς προσπαθούμε εδώ να κάνουμε μία αντικειμενική ανάλυση έτσι ώστε να είμαστε ε, βέβαιοι ότι δεν υπάρχει παραβίαση ουσιοδών ε, κανόνων, όπως ας πούμε ο βασικός κανόνας της προάσπισης ε, μιας βιώσιμης αλληλείας εμείς ε, θεωρούμε ότι υπάρχουν ε, κάποιες βασικές αρχές ε, οι οποίες θα πρέπει να γίνονται σεβαστές και νομίζουμε ότι σε αυτήν την πρόταση γίνονται σεβαστές οι αρχές αυτές και οι κανόνες. Στην δικιά μου εισήγηση, από την άλλη πλευρά, εγώ κράτησα τις δεσμεύσεις μου Ε, λοιπόν, θεωρούμε ότι ε, στην ε, στο δικό μας έγγραφο λέμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει καμία αφαίρεση τμήματων του σώματος επί του σκάφους. Στην πρόταση της Κομισιόν αναφέρεται ότι τα πτερήγια μπορούν να εκφορτωθούν σε, διαφορετικά, σε διαφορετικούς λιμένες και ε, επομένως δηλαδή στην ουσία το σώμα και τα πτερίγια να εκφορτωθούν σε διαφορετικούς λιμένες. Είστε ο Και ε, βεβαίως ε, όταν η εκφόρτωση του σώματος αλλά και των πτερυγίων λαμβάνει χώρα σε διαφορετικούς λιμένες, τότε να καταγράφονται ορθώς αυτές οι εκφορτώσεις. δεν μπορούμε να ε, ε, ε, καταγράψουμε σωστά αυτά τα στοιχεία και δεν έχουμε και αποδείξεις σχετικά με το κατά πόσον γίνεται εξαγωγή μετά την εκφόρτωση. Θα πρέπει να γίνεται ταυτόχρονη εκφόρτωση, εκφόρτωση του σώματος και των πτερυγίων. Ταυτόχρονη εκφόρτωση, εκφόρτωση στο ίδιο λιμάνι λοιπόν. Πώς μπορούμε όμως να βεβαιωθούμε ότι ο έλεγχος, η επιθεώρηση είναι σωστή. Αυτό ε, ρωτήσαμε. Δηλαδή πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι το σώμα και τα πτερίγια τα οποία εκφορτώνονται ανήκουν στο ίδιο, ε, στον ίδιο καρχαρία. Ε, εδώ προκύπτουν ε, επιστημονικά ε, ζητήματα. Ξέρετε ότι τα πτερήγια μπορούν να διαφέρουν αναείδος, επομένως θα πρέπει να μπορεί να ελέγξει κανείς κατά πόσον τα πτερήγια ανήκουν στο ίδιο είδος με το σώμα, κατά πόσον τα πτερήγια είναι πλάγια ή κεντρικά κτλ. Ε, και εμείς είπαμε ότι εντάξει να υπάρξουν περαιτέρω έλεγχοι αλλά δεν μπορούν να υπάρχουν διαρκώς επιπλέον ε, ε, κόστη. Οι οργανισμοί επίσης θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι αλλά εάν όπως είπαμε πριν χρηματοδοτούνται οι οργανισμοί ελέγχου από τους πλειοκτήτες πόσο ανεξάρτητοι μπορεί να είναι. Ε, απ' την άλλη πλευρά, αν θέλουμε ελέγχους αλλά δεν θέλουμε να πληρώσουμε, ε, τότε θα πρέπει με κάποιο τρόπο να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία του οργανισμού. Εάν δεν έχουμε ανεξαρτησία, ασφαλισμένη ανεξαρτησία του οργανισμού, ε, τότε θα πρέπει να δεχτούμε ότι δεν είναι ε, ανεξάρτητος και επομένως ε, δεν είναι σωστός και ο έλεγχος που κάνει. Λοιπόν, η πρόταση έχει ήδη προαγγελθεί, αλλά εμείς μέσω του συμβιβασμού που σας είχα προαναγγείλει επίσης προχωρήσαμε ακόμα παραπάνω. Έχουμε τρεις προτάσεις λοιπόν, οι οποίες ε, περιέχουν ε, υποχρεώσεις για τον Ευρωπαϊκό Στόλο. Έχω προβλέψει και κάποιες άλλες πρόνοιες ε, οι οποίες θα καλύψουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για ε, πραγματική βιώσιμη αλληλεία των καρχαριδών. και έτσι ώστε να γίνεται σωστή αξιολόγηση ε, και των ε, αποθεμάτων, των αλληλευτικών αποθεμάτων των καρχαριδών, αλλά και της αλίας τους πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβουμε σοβαρότατα υπόψη μας και τα μελήματα των μη κυβερνητικών οργανώσεων που γνωρίζουν καλά το θέμα ε, και επομένως να διαμορφωθεί ένα σχέδιο δράσης ε, για, τα, για τους καρχαρίες. Εδώ και χρόνια το ζητούμε αυτό, αλλά η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτιμάει να απαγορεύσει πλήρως την αλία του Καρχαρία και των ε, ειδών Καρχαρία, ε, παρά να κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση. Αλλά αυτό δεν είναι δυνατόν να το δεχτούμε. Αυτό ζητώ λοιπόν μέσω των τροπολογιών και επίσης να γίνει ε, αξιολόγηση του συνολικού αριθμού των ε, καρχαριών αναείδος ε, που έχουν αλλιευθεί. Δηλαδή να έχουμε από πλευρά των πλειοκτητών συγκεκριμένα, συγκεκριμένα ποσά και συγκεκριμένα στοιχεία όσον αφορά το κάθε αλλιευμένο είδος, το βάρος του, το είδος του κτλ. Και επίσης μια δειγματοληψία αναείδος. 15% ε, για 15% για παραπάνω από 100 ε, ε, αλλιευμένα είδη και που θα ανεβαίνει σιγά σιγά 25% και μέχρι 50% για πολλά αλλιευμένα είδη. Και εν πάση περιπτώσει, ολοκληρώνω Πρόεδρε, ναι δεν θα αργήσω αλλά είναι σημαντικά αυτά που λέω. Ε, λοιπόν, ε, σε συνεργασία και με τους επιστήμονες να μπορέσουμε ε, να έχουμε ένα σωστό ιστορικό όσον αφορά ε, τις, τους αλλιευτικούς πόρους των καρχαριοειδών προσπάθησα να απαντήσω εις τα μελήματα όλων των εμπλεκομένων φορέων. Ε, δεν θέλησα να ακολουθήσω τον εύκολο δρόμο, ε, δηλαδή είτε τα επιτρέπουμε όλα είτε τα απαγορεύουμε όλα. και ε, επίσης να αποφύγουμε να ζημιωθεί το σύνολο του ευρωπαϊκού στόλου λόγω ε, υποψιών ε, για παράνομο εμπόριο πτερυγίων. Ξεκίνησα την έκθεση χωρίς προκαταλήψεις και προδικασμένες θέσεις και επομένως έτσι προσπάθησα να ολοκληρώσω την εργασία μου, δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αξιολογώντας ε, όλα τα στοιχεία τα οποία είχα στη διάθεσή μου και βεβαίως και μέσω των τροπολογιών θα ολοκληρώσουμε και τη θέση μας. Είναι γεγονός ότι έχουμε αποκλήσεις ε, απόψεων, αλλά λαμβάνοντα υπόψη την κατάσταση θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να προσαρμοστούμε με ανοιχτό μυαλό, λοιπόν εγώ, με πολύ ανοιχτό πνεύμα ε, παρουσίασα την έκθεση και τις ε, τροπολογίες έτσι ώστε ε, με ισορροπημένο τρόπο να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρωμέδα. Ευχαριστώ πολύ. Πολλά πράγματα έχουμε εδώ. Και θα ήθελα να επισημάνω τα πιο σημαντικά. Πρώτον, εγώ κατανοώ τη βούληση της κυρίας Πατράω να καταλήξει σε έναν συμβιβασμό. Αλλά το πρόβλημα βρίσκεται στη ρίζα του ζητήματος. Αναφέρθηκαν τα κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα. Αλλά ποιες είναι οι κοινωνικο-οικονομικές, τουλάχιστον οικονομικές επιπτώσεις για το στόλο. Διότι εμείς είδαμε μερικά νούμερα, τα οποία όμως αλλάζουν ανάλογα με το πλαίσιο και δεν αποδεικνύεται τελικά Ποια είναι η οικονομική επίπτωση στο στόλο. Πριν από μερικούς μήνες λέγαμε ότι ήταν αδύνατον το να ξεφορτώνει κανείς πτερίγια και ε, σφάγια ε, στο, στο ίδιο λιμάνι. Ότι ήταν αδύνατο. Μα άμα δεν ήταν πρόβλημα τότε, τώρα γιατί να αλλάζει. Εμένα τότε ο βιομήχανος βιομήχανοί μου είχαν πει ότι οικονομικά ήταν μια καταστροφή. Τώρα αλλάξατε και λέτε ότι δεν είναι. Λοιπόν, ότι απο... Ωραία, συμφωνούμε. Λοιπόν, αποβίβαση στο ίδιο λιμάνι. Διαφωνώ. Όταν η συνάδελφος λέει ότι η χωριστή αποβίβαση, εκφόρτωση ε, οδηγεί στο φίνινγκ, ε, αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Όχι, Εάν δεν δέσουμε τα πτερίγια στο σφάγιο, τότε ποτέ δεν θα μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι τα πτερίγια ανταποκρίνονται στο συγκεκριμένο σφάγιο και οι επιστήμονες δύσκολα μπορούν να βρουν άκρη. Διότι μετά δεν ξέρουμε και ποια, κομμάτια του, ποια τμήματα του σώματος θα πετάνε από το πλοίο Θα πρέπει λοιπόν εμείς να λέμε εκφόρτωση των ε, κορμιών, των, των σφάγιων, των καρχαριών με παραδίπλα τα, φτε, τα δεμένα τα Τώρα, για όταν, ε, μιλάμε εμείς, ε, όταν δεν μιλάμε εμείς για τα πλοία με ψυγείο κατάψυξη, δύσκολα μπορούμε να, να, λύσουμε το πρόβλημα, διότι όλο αυτό το εμπόριο γίνεται από πλοία καταψύχτες. Ένα άλλο σημαντικό σημείο για τις μελέτες επιπτώσεων. Λένε πολλά πράγματα. Και είναι σημαντικό να θυμίσουμε ότι αυτό το οποίο λένε είναι να έχουμε αυτό το fish reaming attach option. Να έχουμε δηλαδή την επιλογή να παραμένουν τα φυσική συνοχή με το σώμα. Για τον έλεγχο. Συμφωνούμε απόλυτα ότι χρειάζεται περισσότερος έλεγχος, αλλά έχουμε δύο προβλήματα. Εάν με δυσκολία σήμερα μπορούμε να ελέγξουμε το 5% και το κάνουμε 14% πάλι πολύπλοκο θα είναι. Μόνο δηλαδή το θέμα της διατήρησης των ποσοστώσεων είναι προβληματικό. Και έχουμε και τεράστια βεβαιότητα για το πώς, ε, πού και πώς θα κάνει τον έλεγχο. Τώρα αυτός ο ανεξάρτητος οργανισμός που θα ελέγχει αυτή την δραστηριότητα έχει δύο προβλήματα. Πρώτον, κάποιος πρέπει να τον πληρώσει τον έλεγχο και εγώ δεν έχω καμία εμπιστοσύνη ενός οργανισμού που θα πληρώνεται από τη βιομηχανία για να ε, ελέγχει τη βιομηχανία. Και αν ο έλεγχος γίνεται όπως σήμερα στα λιμάνια, τότε το έχουμε εγγυημένο ότι έλεγχος δεν θα γίνεται. Εξού λοιπόν παραμένουν και όλα τα ζητούμενα ε, που πρέπει να λύσουμε ε, και για την Κομισιόν δηλαδή ε, παραμένουν όλα αυτά ανοιχτά. Εμείς θα κάνουμε τροπολογίες προς δύο κατευθύνσεις. Αυτές της κυρίας Πατράων που υπάρχει δυνατότητα αυτές που δίνουν ε, λύσει το κόψιμο των πτερυγίων δεν θα τις δεχτούμε με τίποτα. Θέλουμε λοιπόν εμείς ε, να τα ξεφορτώνουμε, τα, τους, να ξεφορτώνουμε τους καρχαρίες με τα πτερίγια σε φυσική συνοχή με το χρώμα. Έχουμε τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, έχουμε τις IUCN που μιλάνε για τη διαχείριση των στόκ και όχι μόνο για τον πλετόνο, αλλά για πάρα πολλά είδη τα οποία ε, πλήττονται. Και αναφέρθηκε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για το θέμα της εκφόρτωσης των σφάγιων των καρχαριών με τα πτερίγια σε φυσική συνοχή. Καταλαβαίνω ότι η κυρία Πατράων Ιέβες προσπαθεί να μας πείσει αλλά θέλω να ξέρει για τη δική μας την ομάδα τουλάχιστον είναι ένα θέμα αρχών. Είναι πάρα πολύ εύκολο να λυθεί. Και τώρα όλα αυτά, όλες αυτές οι λύσεις να μπερδεύουμε δηλαδή την κατάσταση από μόνοι μας δεν λύνουν το πρόβλημα αλλά το μπερδεύουν ακόμη παραπάνω. Η κυρία Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με συγχωρείτε, δεν αναγνώρισα το όνομά μου, όπως το προφέρατε. Μάλλον θα το πρόφερα λάθος το λέει ο Ευχαριστώ πολύ την συγκεκριμένη την εκθεσή τη. Έχω κάποιες παρατηρήσεις μόνο. Με ενδιαφέρον παρακολουθώ ότι αναγνωρίζει την ύπαρξη αυτής τη μονάδας αξιολόγησης ε, αντικτύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά πρώτα απ' όλα καθήκον αυτής της ομάδας είναι να αξιολογεί τις δικές μας τροπολογίες, τι είδους επιπτώσεις οι αντικτύπου μπορεί να έχουν και όχι να προσπαθεί να διορθώσει την αντίστοιχη μελέτη που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν λοιπόν πρέπει να γίνει αξιολόγηση του αντικτύπου των τροπολογιών μα, πάλι θα ήταν δύσκολο για τη μονάδα αυτή να κάνει τη δουλειά τη, γιατί θα ήταν πολύ δύσκολο να προβεί σε οικονομική αξιολόγηση κοινωνικο-οικονομικών στοιχείων, θα ήταν ακόμα δηλαδή δύσκολο αυτή η δουλειά. Και πάλι θα ταλαιπωρούνταν με τι εκθέσει τη εισηγητρία, με τι τροπολογίε τη εισηγητρία, όσο και με την έκθεση τη Επιτροπή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ίσω να είναι χρήσιμη αυτή η ομάδα, η μονάδα και θα ήθελα να διατυπώσω την παρατήρηση χωρίς να ξέρω αν τυχόν κάτι ε, έγινε λάθος στη μετάφραση. Έγινε λόγος για μια εύκολη λύση, ε, ότι δεν πρέπει να ψάχνουμε την εύκολη λύση σαν να είναι αυτό κακό πράγμα. Μα ίσως να είναι η πρώτη φορά που μπορούμε να έχουμε μια εύκολη, δηλαδή απλή λύση, η απλή στην εφαρμογή της. Γιατί λοιπόν να είναι κακό και να πρέπει να το αποφεύγουμε. Εγώ νομίζω ότι είναι μάλλον ε, θετικός όρος και όχι αρνητικός όρος, εύκολη είναι προκειμένου, εύκολη λύση. Επίσης, ως προς την δυσκολία καταγραφής των εκφορτώσεων είτε στον ίδιο σε διαφορετικούς λιμένες του σώματος και των πτυριγίων χωριστά. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με την εκφόρτωση του πτυριγίου πάνω στο σώμα, δηλαδή να μην έχει γίνει αποκοπή. Με αυτό λύνουμε το πρόβλημα. Θα πρέπει να Θεωρηστεί αυτό μόνο σαν δυνατότητα στην ε, κοπή, ε, αποκοπή του πτερυγίου στα σκάφη με εξοπλισμό κατάψυξης με πολύ χαμηλό αντίκτυπο. Και έτσι δεν καταλαβαίνω τι διαφορά μπορεί να έχει αυτό, αφού είναι τόσο περιορισμένο ο αριθμό των σκαφών. Αυτή είναι η παρατήρησή μου. Ελπίζω να να σα αφήσει. Παρακαλώ, κύριος Ντέιβις. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εάν ήμουν Ισπανός ή Πορτογάλος ψαράς και δραστηριοποιήμουν στη δραστηριότητα αυτή, θα έλεγα ότι με περηφάνεια με εκπροσωπεί η Μαρία, με υπερηφάνεια βλέπω ότι ε, λαμβάνει υπόψη τις διάφορες απόψεις που διατυπώνονται και δραστηριοποιημουν στην δραστηριοτητα αυτη θα ελεγα οτι με υπερηφανεια με εκπροσωπει η μαρια με υπερηφανεια βλεπω οτι λαμβανει υποψη τις διαφορες αποψεις που διατυπωνονται και προσπαθει να βρει μια λύση που να ικανοποιεί τους πάντες. Κάνει καταπληκτική δουλειά Κοιτάω λοιπόν αυτά που έχει προτείνει εδώ. Πρέπει το, το σώμα να εκφορτώνεται μαζί με το πτερίγιο στον ίδιο λιμένα. Το σκάφος, ο ιδιοκτήτης πρέπει να καταβάλει το τέλος, το, το κόστος της επιθεώρησης. Μπορούμε να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες, αλλά η πρόταση υπάρχει. Τα δεδομένα, πρέπει να συλλέγονται δεδομένα. Πρέπει ο ΛΙΕΑΣ, εφόσον εμπλέκεται στη συλλέγει δεδομένων, και να τα προσφέρει ε, ποσοστώσεις ενδεχομένως ε, να εφαρμόζονται για τους καρχαρίες. Όλα αυτά λοιπόν με στόχο την ε, επίτευξη της, ε, ε, του τελικού μας σκοπού, δηλαδή την προστασία του ή την αποφύγη της μείωσης των αποθεμάτων καρχαρία. Και σε αυτό πρέπει να εξασφαλίσουμε τη σύμπραξη των αλλιέων, έτσι δεν είναι και, είναι και καλό πράγμα, δεν πρέπει να είναι κακό. Πολλά θετικά στοιχεία να έχει η συγγήτρια μου ζήτησε να πάμε μαζί έξω να μου εξηγήσει τα σχέδιά τη, μου εξήγησε τα επιχειρηματά τη. πάρα πολύ καλά, πολύ καλά σχεδόν, σχεδόν με έχει πείσει. Αλλά, αλλά τελικά η ουσία είναι αυτό που ακούστηκε νωρίτερα στην αρχή, το κόστος δηλαδή. Τροπολογία υπάρχει μόνο 8. Το λέει ξεκάθαρα νομίζω, αν βρω το κείμενο τροπολογία 8 όπου λέει ότι θα τα καταφέρουμε αυτά για να αποφύγουμε τις σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές απώλειες για το τομέα που θα προξενούσε η απαγόρευση της εκφόρτωσης ε, ε, σώματος και πτεργίου. Έχω αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι το εξή, ότι ε, εν πάση περιπτώσει έχουμε έναν καρχαρία, τον έχουμε πιάσει, παίρνουμε ένα μαχαίρι, το κόβουμε το πτερίγιο, τον βάζουμε στην κατάψυξη. Πού είναι η απώλεια ακριβώς. Πού είναι η απώλεια. Καταλαβαίνω ότι μπορεί κάποιοι να ενοχλούνται, αλλά σε τι χάνουμε κοινωνικο-οικονομικά, αυτό είναι που δεν αντιλαμβάνομαι. Και αν δεν μπορούμε να πιστούμε για αυτό το επιχείρημα, καταραίει ολόκληρο το οικοδόμημα η Επιτροπή. Για πολύ καιρό προσπάθησε να μα εξηγήσει ότι πρέπει ο Καρχαντή να διατηρεί το πτερυγιό του, κάτι το οποίο και εμεί είχαμε προσπαθήσει να πείσουμε ε, σε προηγούμενα κοινοβούλια και την Επιτροπή. Του πείσαμε εν τέλει. Και θα την ακολουθήσω παρά, παρά την καταπληκτική και λαμπρή δουλειά που έκανε η συγγετρία. Ευχαριστώ κυρία Λόβιν. Ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ ιδιαίτερα την συγγετρία Μαρία, ιδιαίτερα σημειώνω τις τελικές σου, τις καταληκτικές σου παρατηρήσεις, ότι θα πρέπει, όπως είπες, να διατηρούμε πνεύμα ανοιχτό, να προσαρμοζόμαστε στην πραγματικότητα. Και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή πρέπει να αναγνωρίσει ότι κράτη όπως η Κωνσταντίνα, η Ταϊβάνα, έχουν ήδη εισαγάγει τον κανόνα για την ε, μη αποκοπή του πτερυγίου. Υπάρχουν κάποιες άλλες χώρες που σκοπεύουν να τον εισαγάγουν. Είναι κάτι δηλαδή, το οποίο αποτελεί μια τάση ανά τον κόσμο. Την προηγούμενη εβδομάδα η, δημοκρατία, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει να σερβίρεται πλέον σε επίσημο δείπνο πουθενά σούπα πτερυγίου καρχαρία, πράγμα το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό σημάδι μήνυμα ότι ελπίζουμε, αν όχι στο εγγύς μέλλον, πάντως κάποια στιγμή να, μπει να, να μείνει στην ιστορία, να γίνει παρελθόν το ε, πτερίγιο Καρχαρία. Και ασφαλώς θα πρέπει να προσαρμοστούμε όλοι στην πραγματικότητα. Κάποιες από τις λεπτομέρειες που πρότεινες, μου φαίνεται ότι ακολουθούν τελείως εσφαλμένη προσέγγιση και κατεύθυνση. Αναφέρει σε παραδείγματι ένα ποσοστό 14% του πτεργίου σε σχέση με το ε, βάρος του κρέατος, ενώ ε, ε, οι Ηνωμένε Πολιτείες εδώ και πέντε χρόνια τουλάχιστον έχουν 5%. Γιατί να πάμε τόσο πίσω εμείς, γιατί να πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο πίσω, θα ήταν τροπή να το κάνουμε αυτό. Και νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ σοβαρή και απλή λύση, καλή λύση, δηλαδή η εκφόρτωση να γίνεται καρχαρίας και πτερίγιο μαζί, να μην έχει αποκοπεί το πτερίγιο δηλαδή. Και το είπα ε, στο παρελθόν ότι με έχει πλησιάσει και η ισπανική, ο ισπανικός κλάδος που για πολύ μεγάλο διάστημα μου όπως μου εξηγήσει ότι δεν μπορεί να εκφορτώσει το ε, πτερίγιο μαζί με το ε, σώμα, με το σφάγιο του Καρχαρία, γιατί μου λέγανε ότι δεν είναι δυνατόν πρακτικά να γίνει αυτό στον ίδιο λιμένα. Το, το και ο συνάδελφο νωρίτερα. Εν πάση περιπτώσει μετά αλλάξανε την ε, ιστορία τους και τα επιχειρηματά τους, προσπαθούσαν να εξηγήσουν οικονομικές απώλειες και δεν ξέρω τι άλλο. Άρα όλα γίνονται. Ο κύριος Αρσένης. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πιστεύω, διερωτώ με μάλλον, εάν ε, μήπως χρειαστεί να κάνουμε και μια ανάλυση κόστος αποτελέσματος ε, για την απαγόρευση της ε, του δουλεμπορίου. Ξέρετε ότι υπήρξε κάποτε αυτό το φαινόμενο και μετά σταμάτησε. Και παλιότερα επίσης γινόταν η η, να, να ψαρεύουν τεράστια κήτη μέσα στη θάλασσα, να του αποκόπτουν το πρετηρίο και μετά το σφάγιο να ξαναδορίχνεται στη θάλασσα. Ε, ο άνθρωπος απάντησε κάποια στιγμή να σταματήσει το δουλεμπόριο, έτσι μπορεί και να σταματήσει να αποκόπτει το πτερίγιο του Καρχαρία. Το φίνιγμα όπως ονομάζεται. Είπε και η συνάδελφος ότι 25 κράτη-μέλη ήδη έχουν σταματήσει την αποκοπή του πτεριγίου από τον Καρχαρία χωρίς να δεχθούν καμία εξαίρεση ως προς την πλήρη απαγόρευση του ε, της δραστηριότητας αυτής. Έχουν αποφασίσει να εκφορτώνεται ολόκληρο το σώμα του καρχαρίου, ολόκληρο το σφάγιο με το πτυρίγιο δηλαδή μαζί. Οι Ηνωμένε Πολιτείε το ίδιο. Ακόμη και οκτώ χώρες, ε, Μπελιζέ, Κωνσταντίνα, Σαν Σαλβαντόρ, ε, Γουατεμάλα, Ονδούρας, Παναμάς και Κανή δημοκρατία έχουν αποφασίσει να το κάνουν. Ο Παναμά που τόσε φορέ έχουμε κατηγορήσει, η Ταϊβάν που τόσε φορέ έχουμε κατηγορήσει για την αποκοπή του πτερυγίου, πρόσφατα την απαγόρευσε. Και φαίνεται να προχωρεί προς αυτή την πολιτική του να εκφορτώνεται το σφάγιο ολόκληρο με το πτερίγιο στη ράχη. Άρα το μόνο λογικό πράγμα που μπορεί να κάνει κανείς είναι να απαλληφθεί το άρθρο 4, να καταργηθεί η παρέκκληση και η αδίποτε παρέκκληση. Η κυρία Νέβες με την οποία είχαμε πολύ καλή συνεργασία σε όλη τη διαδικασία με την οποία προσπαθήσαμε να δούμε κάθε επιχείρημα εις βάθος ε, και να ε, συζητήσουμε ουσιαστικά. Μας λέει ότι η λύση θα ήταν να περιοριστεί η πρόταση σε μία παρέκκληση μόνο για με τα σκάφη, στα σκάφη με εξοπλισμό κατάψυξης. Εγώ το κοίταξα αυτό. Μα μόνο σκάφη με εξοπλισμό κατάψυξης προβαίνουν σε αυτή την πρακτική πλέον. Άρα δεν μου λέει τίποτα καινούριο. Στην ε, μελέτη αντικτύπου, ξέρετε ότι υπάρχει μελέτη αντικτύπου για την πρόταση αυτή, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα που έχουν διεξοδικά μελετηθεί. Το πρόγραμμα δράσης ε, για τον ε, Καρχαρία υιοθετήθηκε το 2008. Η ιδέα της εκφόρτωσης σφαγίου μαζί με, τον, ε, με το πτερίγιο στο ίδιο, στον ίδιο λιμένα, ξέρετε, έχει ζητηθεί. Έχει αναλυθεί. Αλλά ξέρετε, λόγω του ποσοστού, λόγω του τρόπου με τον οποίο έχει διατυπωθεί αυτή η αναλογία, είναι πολύ εύκολες οι απάτες. Είναι εύκολο δηλαδή να ψαρέψει κανείς αυτό το κήτος, να του αποκόψει, να αποκόψει τα για δύο καρχαριών και να καταγράψει το ίδιο βάρος πτεριγίου για δύο, για έναν καρχαρί αντί για δύο και έτσι να κερδίσει αντίστοιχα τον χώρο που προβλέπεται. Και ξέρουμε ότι το πρόβλημα είναι ήδη εντοπισμένο σε περίπτωση, στην περίπτωση της ε, Ισπανίας στους χώρους 8 και 9 ήδη. Και ούτω ή άλλω, ακόμη και να δεχόμαστε αυτή την αρχή, είναι, την παρέκκληση, είναι πολύ ασαφή η κατάσταση. Πώ διαφορετικά είδη καρχαριών μπορεί να έχουν διαφορετική αναλογία πτερυγίου σώματο. Όπω άλλωστε και άλλοι συνάδελφοι εξέθεσαν. η πρόταση ο αρμόδιος, ο υπεύθυνος για το σκάφος με εξοπλισμό κατάψυξης να, ε, να έχει την ευθύνη για την επιθεώρηση που θα γίνει κατά την εκφόρτωση. Και πάλι θα ρωτήσω τι είδους ε, αντίκτυπο μπορεί να έχει αυτό το μέτρο ανάλυση κόστου αποτελέσματος δηλαδή. Αλλά θα πω και το εξή. Πώς είναι δυνατόν εγώ να ελέγχω από κάποιον τον οποίο εγώ πληρώνω, εγώ αμείβω. Μπορεί και σε έναν ιδεώδη κόσμο να το καταφέρουμε και αυτό, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο ιδεατό. Και θα ήθελα να δηλώσω κάτι το οποίο θεωρώ θεμελιώδες, κλείνοντας πρόεδρε. Το να παραμένει το πτέρυγιο πάνω στο ζώο είναι η απέτηση που έχει διατυπώσει η κοινή γνώμη μέσω της γενικής διαβούλευσης. Είναι σαφές αυτό. Είναι αυτό το οποίο ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη γραπτή του δήλωση, με 450 υπογραφές. Και επίσης τα κράτη-μέλη, 27 με πλειοψηφία 25 κρατών μελών, ζήτησαν το ίδιο πράγμα. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει συχνά. Δηλαδή, είναι δυνατόν εμείς να είμαστε λιγότερο φιλόδοξοι από την Επιτροπή, από το Συμβούλιο, από τους πολίτες και να υπολοιπόμεθα και τη κοινή λογική. Δεν νομίζω. Ευχαριστώ, κύριο Σάντσε εγώ άκουσα με ιδιαίτερο σεβασμό όλες τις θέσεις και από την πρώτη στιγμή θα πω ότι εγώ είμαι κοντά στην κυρία πατράω. Δεν μιλάμε ούτε για βιοπικιλότητα ούτε για υφοροαλία, όλοι συμφωνούμε. Υπάρχει μια κοινότητα στη Γαλλικία που έχει, πολύ σημαντική, που έχει σημαντική δραστηριότητα σε αυτόν τον τομέα. Στη στην Γαλήθεια σίγουρα δεν θα βρείτε εστιατόριο το οποίο να σας σερβίρει σούπα με πτερίγια χαρχαρία, πολύ πιθανό στη Βαρκελόνη, στη Στοκχόλμη. Να ξέρετε ότι ο στόλος μας ε, αποβιβάζει στον ίδιο λιμένα, εκφορτώνει στον ίδιο λιμένα. Στη χώρα μας το σώμα καταναλώνεται και θα, αυτό θα το βρείτε ναι στους καταλόγους ε, των εστιατορίων και τα πτερίγια τα στέλνουν στις αγορές που τα καταναλώνουν αυτά τα πτερίγια. Υπάρχει όντως ένα πρόβλημα ελέγχου. Αλλά δεν μπορούμε να μπούμε στην καρικατούρα του Γκρούτσο Μάρξ που λέει ότι η πολυπολιτική έγκυται στο να βρίσκει προβλήματα εκεί όπου δεν υπάρχουν και να τα λύνει δίνοντας λαθεσμένες λύσεις. Και δεν μπορούν να μας λένε ότι οι τομείς, ε, οι κλάδοι οι οποίοι απασχολούνται με αυτήν την αλία ε, δεν ε, ε, ενδιαφέρονται, δεν ξέρουν τη δουλειά τους και δεν ενδιαφέρονται να διασφαλίσουν τους φυσικούς τους πόρους που θα τους συνεχίσουν τη δουλειά τους. Η βιομηχανία γνωρίζει πολύ καλά ότι η φόρμουλα που τους προτείνει ο κανονισμός είναι σωστή και φυσικά αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται και με τον έλεγχο. Ο έλεγχο σίγουρα είναι κόστος, αλλά από την άλλη μεριά είναι και εγγύησης. Και αυτό οδηγεί σε μία λογική γραμμή. Γι' αυτό πιστεύω ότι Μπορεί να πιστεύουμε ότι υπάρχει μία ενιαία λύση για το πρόβλημα, αλλά δεν ξέρουμε, δεν βρήκαμε ποιες είναι οι πιο λογικές αναλλακτικές λύσεις. Ε, αν εμείς πρέπει να εκφορτώνουμε από κοινού, να ξέρετε ότι αυτή η δραστηριότητα που προτείνεται εδώ θέλει αύξηση κόστους διότι ορισμένοι θα κάθονται και ορισμένοι θα δουλεύουν. Αλλά άμα όμως εκφορτώνονται χωριστά τα δύο τμήματα, ξέρετε με τους δορυφόρους μπορούμε κάλλιστα να δούμε μέχρι το τελευταίο μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια της εκφόρτωσης. Το μόνο που κάνουμε εδώ όμως εμείς είναι να ρυθμίζουμε με επιθετικό τρόπο, διότι δεν έχει κανένα νόημα. Είτε εκφορτώνονται σφάγια και πτερίγια σε ένα λιμάνι, είτε σε δύο. Είμαι κατά του φίνινγκ, είμαι υπέρ του ελέγχου, θέλω μέτρα πραγματικού ελέγχου διότι εγώ θεωρώ παράλογο να τιμωρούμε έναν τομέα, έναν κλάδο και παράλληλα να τιμωρούμε και όλους τους καταναλωτές. Η κυρία Πράγα. Φράγα. Εγώ θα πω ότι το πιο εύκολο για την κυρία Πατράου θα ήταν να υποστηρίξει ή να φέρει αντιρρήσεις στην ευρωπαϊκή πρόταση. Εγώ πιστεύω ότι το σημαντικό εδώ ήταν να βρούμε μαζί με τον κλάδο ποιες είναι οι καλύτερες συμβιβαστικές λύσεις που θα... Και για τους ίδιους δηλαδή και για τον κλάδο, και για τον οποίο κλάδο επίσης αυξάνεται το κόστος. Να ξέρετε ότι με αυτά που μας λέτε, ο στόλος θα χάσει πάρα πολλά. και είναι έτοιμοι να πληρώσουν ποσά τα οποία ρωτώντας τον οργανισμό Βέριτα 6 με 10.000 δολάρια αναπλοίο στη θάλασσα. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος ε, του εχειρήματος της Κομισιόν Και αυτό το κόστος λειτουργεί προς, προσθετικά. Εμείς λοιπόν ψαρεύουμε τον καρχαρία, μετά χωρίζουμε τα πτερίγια, τυλίγουμε σε ένα δίκτυ και Ξέρετε ότι αυτό δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό το οποίο συνηθίζεται, διότι σύμφωνα με τον έτρο θα πρέπει τα δίχτυα να ξαπέφτουν στη θάλασσα. Να ξετυλίγονται, συγγνώμη. Έχουμε και απώλεια ποιότητα, διότι αυτή τη στιγμή εκφορτώνονται αυτοί οι καρχαρίες. Θα πρέπει εκεί, στο λιμάνι, να κόψουμε εντελώς τα χαραγμένα πάνω στο σώμα πτερίγια, και χάνουν την προέλευση. Και όλα αυτά γίνανε με έναν τρόπο ιδιαίτερα αναλυτικό και πρέπει να βοηθήσουμε εμείς την κυρία Πατράο. Εμείς μπορέσαμε να επαληθεύσουμε όλα αυτά τα πράγματα συνεργαζόμενοι με τον κλάδο. Πρέπει να δούμε που εργάζονται επίσης στη Μαδαγασκάρη, στο Πράσινο Ακροτήρι. και ο έλεγχος μπορεί να είναι ιδιαίτερα ελαστικός σε αυτά τα μέρη. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να καταλήξουμε σε αυτά, στο συμβιβασμό που μας προτείνει η κυρία ε, Πατράο. και να ακούσουμε τέλος πάντων τους επιστήμονες, διότι οι επιστήμονες είναι αυτοί που ξέρουν τα πράγματα και όχι εμείς, και να εξετάσουμε αναλυτικά και να σας στείλω και όλα τα στοιχεία που θέλετε, ούτω ώστε όλοι να λάβουν την απόφασή τους κόγκιτο κάουσα. Αλλά πρέπει να προχωρήσει όλη αυτή η ιστορία γιατί και μεγάλες προσπάθειες καταβάλαμε και ένα σωρό χρόνο χάσαμε και θέλουμε να έχουμε καλύτερη αλία. Ευχαριστώ κυρία Φράγα. Από την Κομισιό. Η Επιτροπή παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ξεκινώ και εγώ ευχαριστώντας την εισηγητρία για τη δουλειά της και τις προσπάθειες για αναζήτηση συμβιβαστικών λύσεων. Καθώς επίσης και μια πολύ καλή προσπάθεια για μια έκθεση ισόρροπη, ουδέτερη. Για την προσπάθεια να καταγράψει τις ε, θέσεις όλων των εμπλεκομένων. Πρέπει να επισημάνω ότι η Επιτροπή προσπάθησε να κάνει το ίδιο και εμείς είχαμε εντατικές διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες, με κυβερνητικές οργανώσεις, τον τομέα, της ε, κυβερνήσεις, των κρατών και αυτό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τόσο κατά τη διάρκεια της περίοδου διαβουλεύσεων, όσο και πριν, μετά και κατά τη διάρκεια των διαφόρων βημάτων που αφορούν την αξιολόγηση αντικτύπων. Και έτσι φτάνω στην παρατήρησή μου, τη σχετική με την ποιότητα της ε, μελέτης αντικτύπου. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να δηλώσω, όπως έχω πράξει και στο παρελθόν, ότι δώσαμε τη δυνατότητα στον τομέα να μας δώσει κάθε είδους δεδομένα, ποσοτικά, ποιοτικά, πρακτικές πληροφορίες και το καθεξής, για μια περίοδο που ξεπέρασε τα δύο χρόνια. Δεδομένα τα οποία εισέρευσαν, λάβαμε πολλά χρήσιμα δεδομένα από τον τομέα, πάντοτε δεν τυπώναμε επερωτήσει, λαμβάναμε περαιτέρω πληροφορίες και δεδομένα. Δυστυχώ, τα ποσοτικά δεδομένα, τα δεδομένα τα οποία εν μέρη ανέφερε σήμερα παραδείγματι η κυρία Φράγα, τα στοιχεία τα σχετικά με το επιπλέον κόστος ανασκάφους και το καθεξής, τα λάβαμε από τον τομέα μόνο τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά αμέσως μόλις τα λάβαμε με τη μορφή πινάκων από τους εκπροσώπους του τομέα. Δώσαμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε μαζί τους, να αναλύσουμε τα δεδομένα, γιατί ήταν πολλά τα ερωτηματικά. Και έτσι είχαν ακόμα την ευκαιρία μερικές εβδομάδες αργότερα να μας δώσουν νέες πληροφορίες, ανάλυση κόστους και θα αναφερθώ και στο κόστος της αρπιγέρα όπως ονομάζεται του ειδικού καλύματος που χρησιμοποιείται για την προστασία του σφαγίου του Καρχαρία και επίσης τη διαδικασία που μας εξήξαν τη διαδικασία που ακολουθείται για, την, για τον Καρχαρία μετά την κατάψυξη. Παρακολουθήσαμε βίντεο, είδαμε πάρα πολλές εικόνες, φωτογραφίες που μας έδωσε ο τομέας, ο κλάδος. Μαζί τους αναλύσαμε όλη τη διαδικασία της κατάψυξης, της εκφόρτωσης, της αφαίρεσης του πτερεγίου, της αποκοπής του πτερεγίου μετά την κατάψυξη και συμπεράναμε και συμφωνεί και ο κλάδος ότι υπάρχει ο εκπρόσωπος του κλάδου με τον οποίο συζήτησα εγώ, ο κύριος Χαβί Καράτ, μου είπε ότι συμφωνεί πως υπάρχει περιθώριο σημαντικό για βελτίωση των τεχνικών που χρησιμοποιούνται, που θα οδηγούσε και σε βελτίωση σημαντικού του κόστους. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό το σημαντικό σημαντική δεν το γνωρίζω, ούτε μπόρεσε ο κλάδος να μου δώσει μέχρι τώρα κάποιες επαρκείς πληροφορίες. θα περάσουμε στις ε, ταυτόχρονες εκφορτώσεις. Μπορεί να υπάρξει βελτίωση ως προς το status quo, αλλά οι ταυτόχρονες εκφορτώσεις ένα λιμόνι, εφόσον υπάρχει αποκοπή δηλαδή του πτερυγίου, από το σώμα δεν σώζει, δεν επιλύει πολλά από τα προβλήματα που έχουμε και επί παραδείγματι δεν επιλύει το ζήτημα της αναλογίας ε, ε, ως προς το βάρος γιατί πρέπει να εφαρμοστεί το καθεστώς αναλογίας επί του βάρους για να ξέρουμε ότι δεν έχει γίνει ε, παράνομο φίνινγκ, ότι δεν έχει δηλαδή απορριφθεί στη θάλασσα το σώμα του καρχαρία. Μπορεί να διευκολύνεται ο έλεγχος στην ταυτόχρονη εκφόρηση αλλά πάντως δεν εγγυάται την, ότι αποτρέπουμε ουσιαστικά το φίνινγκ. Υπήρχε επίσης ένα ζήτημα ως προς απαγορευμένα είδη που έχουν πτερίγιο πολύ πιο πολύτιμο από αυτό των μη απαγορευμένων για την αλία ψαριών, ε, καρχαριών συγκεκριμένα. Και έτσι βλέπουμε ότι υπάρχει ο κίνδυνος να αλλιεύονται αυτοί οι πολύτιμοι καρχαρίες, ε, να αφαιρείται το ε, πτερήγιό τους και να απορρίπτουν αυτή τη θάλασσα. Εμεί θέλουμε να αποτρέψουμε ακριβώς αυτό με την ε, εκφόρτωση του σώματος ολόκληρου μαζί με το πτερήγιο. Η κυρία Πατράου Νέβες έχει κάνει λοιπόν την προσπάθειά της και προτείνει ενισχυμένους ελέγχους. Συμφωνούμε σε αυτό. Πιστεύουμε ο τρόπος να ενισχυθεί ο έλεγχος με χαμηλότερο κόστος είναι να παραμείνει το πτερίγιο πάνω στο σώμα του καρχαρίου. Και έτσι η πρόταση για την πρόσληψη ανεξάρτητων σωμάτων ε, που θα διεξήγαγαν τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις με προβληματίζει ως προς τη λέξη ανεξάρτητα. Όταν ε, μέσα στην ίδια φράση βλέπουμε προσλαμβάνονται από τον κλάδο. Εδώ βλέπω μια αντίφαση. Δεν αντιλαμβάνομαι πώς μπορεί κάποιος τον οποίο, έχω προσλάβει να μην έχει ε, σύγκρουση συμφερόντων ως τον έλεγχο που θα μου κάνει. Αυτά είχα να πω, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Για να ολοκληρώνουμε, η κυρία Πατράου έχει το λόγο. Πολύ σύντομα παρακαλώ όμως, ε. Βεβαίως, Πρόεδρε, θα είμαι πανσύντομη. Για καθένα από αυτά τα σημεία... Θα ξεκινήσω με την Κομισιόν. Μεγάλη μου χαρά πάντα να την ακούω, εκπλήσωμε όταν λέει ότι είναι αντιφατικό να λέμε ότι ο, ε, να χρησιμοποιούμε τον όρο ανεξάρτητος. Μα η Κομισιόν είναι αυτή που χρησιμοποιεί τον όρο ανεξάρτητος οργανισμός και σε πάση περιπτώσει οι ανεξάρτητοι οργανισμοί λειτουργούν για τα άλλα ψάρια γιατί για τους καρχαρίες δεν πρέπει να δουλέψουν. Τώρα συμβιβαστική πρόταση, εγώ είμαι αυτή που την, ε, που την παρουσιάζω. Η Κομισιόν τι έκανε δύο χρόνια, πλάκα έκανε, χρόνο έχανε. Πέρασαν δύο χρόνια χωρίς κανένα συμβιβασμό. Και ο κλάδος δεν πρέπει να κάνει αυτή τη δική σας δουλειά. Εσείς πρέπει να κάνετε τη δική σας. Δεν είναι ο κλάδος που πρέπει να σας παρέχει τα στοιχεία. Εσείς πρέπει να τα μαζεύετε και να είναι αξιόπιστα. Αγαπητοί συνάδελφοι, όλη αυτή η ιστορία της ε, μελέτης επίπτωσης Εμείς ε, την έχουμε κάνει και είναι μελέτη της επίπτωσης της επίπτωσης ε, της, επίπτωσης της Κομισιόν που η Κομισιόν έρχεται και μας λέει ότι δεν κάναμε. Και αν η Κομισιόν εργάστηκε τόσο στενά με τον κλάδο ε, και έχουν μαζέψει όλα αυτά τα άπειρα στοιχεία και τα έχουν μαζέψει και δέκα φορές, μα που είναι γιατί δεν μας τα έδωσαν. Μετά η Κομισιόν μας λέει ότι η ταυτόχρονη αποβίβαση δεν λύνει το πρόβλημα. Αλλά εγώ διάβασα και τι έλεγε και η Επίτροπος πριν από καιρό και έλεγε ότι το πρόβλημα είναι η έλλειψη ταυτόχρονης ε, αποβίβασης. Ε, λοιπόν, η Κομισιόν τι κάνει. Μία μέρα λέει το ένα πράγμα και την άλλη μέρα λέει το άλλο. Ειλικρινά δηλαδή ε, και γραπτά πια λέγεται ότι, ότι υπάρχει ταυτόχρονη εκφόρτωση Ε, σφάγιου και πτερυγίων, τότε έχουμε το πρόβλημα του σπίνινγκ. Λοιπόν, αυτοί που έπρεπε να παρουσιάσουν το πρόβλημα δεν το παρουσιάσανε, την πρόταση συγγνώμη δεν το παρουσιάσανε. Κυρία Γκέρλινγκ, με καταλάβατε, ωραία δεν πρόφερα το όνομά σας ε, τόσο άσχημα. Εσείς υποστηρίζετε ότι είναι περίεργο που άσκησα κριτική σε αυτό το, στον επιθετικό προσδιορισμό απλό. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι δική μου δουλειά να, να ψάχνω απλές λύσεις. Εγώ πιστεύω ότι η ευθύνη μου είναι μετά από την ακρόαση όλων των ενδιαφερομένων να βρω τη λύση που δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητα η πιο απλή, αλλά η καλύτερη και που θα παντρεύει τις θέσεις όλων. Εκτίμησε ιδιαίτερα την τοποθέτηση της συναδέρφου Λέβιν όταν λέει ότι ο ισπανικός στόλος δεν, δεν έχει κανένα συμφέρον να ξεφορτώνει στο, ίδιο λιμάνι σφάγια και πτερίγια γιατί έχουν διαφορετική, διαφορετικό προορισμό το σφάγιο και τα πτερίγια. Λοιπόν, τώρα δεν μπορεί να είναι και οι δύο καλές, οι λύσεις καλές. Ή η α λύση είναι καλή ή η β είναι καλή. Εμείς, όπως είπε και η Κάρμεν, συνεργαστήκαμε ιδιαίτερα με τον κλάδο. Λοιπόν, Αφήστε τις προκαταλήψεις και τις ε, προκατασκευασμένες ιδέες και εξετάστε αναλυτικά τις προτάσεις. Κάθε φορά το να λέμε τα ίδια και τα ίδια, ε, ειλικρινά, ε, είναι σπατάλι χρόνου. Αυτό ισχύει για όλους μας, δεν το λέω για κάποιον ιδιαίτερα. Λοιπόν, είχαμε λιγότερες πληροφορίες, είχαμε διαφορετικές απόψεις. Τώρα που έχουμε παραπάνω πληροφορίες, ας μην κλείσουμε την πόρτα και ας κοιτάξουμε να κάνουμε σοβαρή δουλειά. Η κυρία Λέβιν λέει ότι στις επίσημες, ε, στα επίσημα δείπνα με τους Κινέζους δεν μας δίνουν σούπα με πτερίλια καρχαρία. Άρα σημαίνει ότι η αγορά έχει αρχίσει και εξαντλείται. Μα ο καρχαρίας, να ξέρετε, χρησιμοποιείται συνολικά, όχι μόνο τα πτερίγια. Και αν στις επίσημες στα επίσημα δείπνα με των Κινέζων δεν θα σερβίρουν σούπα καρχαρία, πτεριγίων καρχαρία. Να ξέρετε ότι το σφάγιο είναι ούτως ή άλλως το πιο αποδοτικό. Και δεν ορίζεται η αγορά από το αν χρησιμοποιούν στα επίσημα δείπνα οι Κινέζοι τα πτερίγια ή όχι. Τώρα, ακούσατε χθε τον Κύπριο Υπουργό, δεν ήξερε καν τι είναι τα πτερίγια και τι είναι οι καρχαρίες, ούτε ήξερε ότι το Κοινοβούλιο συζητάει αυτό το θέμα για την απάνθρωπη πρακτική της αφαίρεσης του πτεριγίου εμείς λοιπόν θα πρέπει να ακούσουμε ένα συμβούλιο το οποίο δεν ξέρει καν γιατί μιλάει. Και αυτό συμβαίνει συχνά και μεταξύ μας. Υπάρχουν χώρες που δεν έχουν καν θάλασσα. Και αυτό ισχύει για όλα τα θέματα, όχι μόνο για αυτό. Έχουμε 27 χώρες που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και όχι απλώς να κάνω αντιπολίτευση λέγοντας εντάξει δεν είναι το δικό μου συμφέρον οπότε ας κουρεύονται οι υπόλοιποι. Υπάρχουν σημεία για τα οποία δεν δόθηκε απάντηση. Κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις. Αυτό γιατί η Κομισιόν δεν έκανε τη δουλειά τους. Εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο κάναμε δουλειά μια χαρά. Το είπαμε και το συζητήσαμε και σε προηγούμενες ανταλλαγές απόψεων. Μετά μας είπανε ότι δεν υπήρξε ανταπόκριση μεταξύ των σφάγιων και των πτερυγίων. Εγώ άκουσα ένα σωρό επιστήμονες και μου είπαν ότι πάρα πολύ εύκολα μπορούμε να βρούμε εμείς ποιο πτερίγιο ανταποκρίνεται και σε ποιον καρχαρία. Οπότε οι καρχαρίες είναι οι ίδιοι. Είτε πρόκειται για, την, ε, για, την, ε, για, το, για το πάνω πτερίγιο ή το κάτω πτερίγιο, Μπορούμε να το βρούμε κάλλιστα. Λοιπόν, εδώ πολλοί είστε επιστήμονες, πράγμα συγχαρητήρια, αλλά ας ακούμε τους εμπειρογνώμονες. Τώρα το ότι δεν αλλάζουν οι όροι για την κατάψυξη ε, στη θάλασσα, ε, κάνετε λάθος. Αλλάζουν πολλά πράγματα και αναφέρετε και την Ταϊβάν, μα είναι άσχετη η Ταϊβάν διότι πρόκειται για στόλους οι οποίοι δεν καταψύχνουν στη θάλασσα, μόνο φρέσκο ψάρι εμπορεύονται. Ο ανεξάρτητος τώρα οργανισμός, εδώ ήδη απάντησα, δεν θέλω να χάσω χρόνο σε αυτό. Πρόεδρε, υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό τώρα και εδώ ολοκληρώνω. Οι ζημιές. Τα, τις περισσότερες από αυτές τις ζημιές τις ανέφερε η Κάρμεν. Γίνεται σπατάλη ενέργειας όταν εμείς ε, ε, έχουμε ψάρι πιο ζεστό και πρέπει να το παγώσουμε αμέσως. Ε, επίσης, ξοδεύουμε και σε εργατικά χέρια για την ψήξη απόψυξη, μετά για το υλικό απόψυξη, απόψυξη και ξανακατάψυξη, σπατάλη ενέργειας, Θα ήθελα λοιπόν να στείλω όλα αυτά τα νούμερα στους συναδέλφους που δεν ε, υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο εδώ δεν το βρήκαμε. Η Κομισιόν μας είπε ότι δεν, υπάρχει τεχνική δυνατότητα για να δούμε ποιο είναι το στόκ των ε, καρχαριών. Εσείς ξεχάστε το σήμερα ότι ο κλάδος θα συνεργαστεί με τους επιστήμονες τώρα. Εγώ θα καταθέσω τροπολογίες. Ε, αν υπάρξουν αν υπάρξουν λύσεις πρέπει να είναι λύσεις με τάκ και με ποσοστώσεις ο κλάδος σίγουρα πρέπει να αλλάξει τη μέθοδο εργασίας αλλά πιστεύω ότι αυτή η πρόταση έκθεσης βοηθάει και στις ανησυχίες του κλάδου. Ευχαριστώ κυρία Πατράου, ευχαριστώ και τους διερμηνείς γιατί ήταν δύσκολη η διερμηνία σήμερα. Και οι διερμηνείς ευχαριστούν τον Πρόεδρο. Στις 18 του μηνός τελειώνει η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών, 12 το μεσημέρι. Σημείο 20. Πρωτόκολλο συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Γουινέας Μπισάου για τις δυνατότητες αλίας και αποζημίωση σχετικά με τη συμφωνία αλίας με τα δύο μέρη είναι ένα θέμα που όπως γνωρίζετε το ανέλαβε επίσης η κυρία Πατράο. Τώρα με το πραξικόπημα κλπ. Η διαδικασία εκκρεμεί και θα θέλαμε απλώς η Κομισιόν να μας πει τα τελευταία και να έχουμε μία μικρή ανταλλαγή απόψεων. Μόνο 20 λεπτά έχουμε για όλα. Κομισιόν έχει το λόγο και παρακαλώ ησυχία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω όντως τη χαρά να σας ε, κάνω μια ε, ενημέρωση όσον αφορά την κατάσταση με τη Γουινέα Μπισάου ε, και τα τεκτενόμενα σχετικά με την ελληνική Συμφωνία με τη χώρα αυτή. Είναι μια συμφωνία που αφορά πολλά είδη, πολύ σημαντική λοιπόν για τον στόλο μας. Έχουμε μια παλιά καλής ποιότητας σχέση παρά τις δύσκολες πολιτικές καταστάσεις ε, της χώρας αυτής. Ε, επίσης είναι μια χώρα η οποία και τώρα ε, διανύει ιδιαίτερα δύσκολη πολιτική κατάσταση. Στις 15 Ιουνίου τρέχοντος έτους εξέπνευσε το πρωτόκολλο συμφωνίας το οποίο ήταν διαρκείας ενός έτους Ιούνιος 2011 Ιούνιος 2012 λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες κατάστασεις, διαπραγμάτευσης υπήρξαν εμπλοκές κλπ. Και γι' αυτό λοιπόν απεφασίστη τότε να έχει ισχύ ενός έτους το πρωτόκολλο. Εν τω μεταξύ υπήρξε πραξικόπημα στην Γουινέα Μπισάου την 12η Απριλίου και επομένως ε, ολοκληρώθηκε και η αλληλεία μετά από μερικές μέρες με την έννοια ότι ε, δώσαμε ε, οδηγία στον ε, στόλο να σταματήσει την αλληλεία τον Απρίλιο του 2012. Κυρίως όταν μάθαμε ότι, υπήρξα, ότι θα υπήρχαν και υλικοί κίνδυνοι ε, για το στόλο μας ε, στα ύδατα της Γουινέας Μπισάου. Ε, γύρω στα μέσα Απριλίου λοιπόν ο στόλος μας στην ουσία απεσήρθη από τα ύδατα της χώρας αυτής. Όσον αφορά το νέο πρωτόκολλο, είχαμε διαπραγματευτεί στην αρχή του χρόνου ένα νέο πρωτόκολλο συμφωνίας αλλιευτικής να πω θα πω δύο λόγια μετά για το περιεχόμενο, να αναφερθώ πρώτα στις διαπραγματεύσεις εμείς ολοκληρώσαμε τις διαπραγματεύσεις μας που πλευρά Εκτελεστική Εκτελεστικής ε, ε, δηλαδή υποβάλαμε τις προτάσεις ε, και στο Συμβούλιο, γνωρίζοντας ότι έχει παγώσει η εξέταση των εν λόγω προτάσεων ε, μέχρι νεοτέρας, μέχρι δηλαδή η πολιτική κατάσταση να βελτιωθεί στη χώρα αυτή μέχρι ότου επανέλθει ε, σε φυσιολογική κατάσταση, ε, αλλά εν να έχουμε ολοκληρώσει τις προτάσεις έτσι ώστε άμεσα να μπορούν να ξαναρχίσουν οι ελευτικές ε, διαδικασίες πληροφορήσαμε τις αρχές της, αρχές της Γουινέας Μπισάο με προφορική ενημέρωση της 13ης Ιουνίου ότι δεν θα υπήρξε επανεκκίνηση των αλλιευτικών ε, διαδικασιών. Ε, είπαμε επίσης ότι δεν θα δεχόμαστε οποιαδήποτε ε, ιδιωτική αδειοδότηση και επομένω, ε, ο αλλιευτικό τόλος, λαμβάνοντα υπόψη τι παρούσε συνθήκε στη Γουινέα Μπισάου, δεν θα μπορούσαν με κανένα τρόπο να αλλιεύσουν στα ύδατα τη Γουινέα Μπισάου. Ε, πάγωσε λοιπόν η εξέταση ε, της ε, πρότασης στο Συμβούλιο μέχρι να βελτιωθεί η πολιτική κατάσταση στη χώρα αυτή. Όσον αφορά το νέο πρωτόκολλο το οποίο διαπραγματευτήκαμε στην αρχή του τρέχοντος έτους, πρέπει να πω το εξή. Ε, είχαμε αρκετά προσπαθήσει να βελτιώσουμε στα πλαίσια του πρωτοκόλου αυτού δύο στοιχεία. Πρώτα απ' όλα την αηφορία και την διακυβέρνηση. Όσον αφορά την αηφορία, τη βιωσιμότητα, πρέπει να υπογραμμίσω ότι μειώσαμε την ε, ικανότητα αλίευσης έτσι ώστε να λάβουμε σοβαρά υπόψη την, υπο... την ε, χρήση ε, και επίσης λάβαμε υπόψη ε, τη γνωμοδότηση της κοινή Επιστημονικής Επιτροπής. Ε, επίσης όσον αφορά την αλληλεία της Γαρίδας λάβαμε υπόψη μας το μέγεθος του βρόχου των δικτυών καθώς επίσης και τα στοιχεία για την, βιολογική, για την αναπαραγωγή του είδους. Επίσης το σύστημα VMS καθώς επίσης και το, την ετήρηση ηλεκτρονική ηλεκτρονικού ημερολογίου του πλοίου. Όσον αφορά τη διακυβέρνηση, έγινε δεχτή από την Γουινέα Μπισάου και ε, ο όρος της ε, αιρεσιμότητας ε, της στήριξης του τομέα, αλλά και η ρήτρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, θελήσαμε να ενδυναμώσουμε την προστιθέμενη αξία αυτής ε, της συμφωνίας για την χώρα και για, τον, ε, για τους πολίτες της Γουινέας Βησάου. Επίσης, προτείναμε και αύξηση της συμβολής των πλειοκτητών. Λοιπόν, η συμφωνία αυτή, η οποία ήταν καλή συμφωνία, αλλά που δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ, είναι παγωμένη αυτή τη στιγμή παρακολουθούμε από κοντά και στενά την πολιτική κατάσταση σε συνεργασία ε, με τους ε, ε, συναδέλφους της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης καθώς επίσης και με τους συναδέλφους της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας Επιτόπου. Περιμένουμε λοιπόν και δεν μπορούμε μέχρι να αρχίσει, μέχρι να διευθετηθεί το πολιτικό ζήτημα, δεν μπορούμε να προωθήσουμε τη συμφωνία αυτή ούτε τη θέσουμε σε Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Πατράου. Θα είμαι σύντομη, Πρόεδρε. Όσον αφορά σε αυτήν τη συμφωνία, εγώ πάντοτε ήμουνα συχνά μάλλον ε, επικριτική γιατί θεωρούσα ότι πάντοτε είχαμε μεγάλη ψηλή συνεισφορά με μικρές ευκαιρίες αλίας. Τώρα για το πρωτόκολλο, αυτό το πρωτόκολλο με τη Γουινέα Μπισάου, ε, καταλαβαίνουμε ότι τα νούμερα είναι διαφορετικά, ε, έχει αυξηθεί η συνεισφορά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα όσον αφορά συνολικά την αλία έχουμε μία ελαφρά αύξηση ε, των αλλιευμάτων, οπότε η αντιστάθμιση για την Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλώνει. Εγώ με ευχαρίστηση μπόρεσα άκουσα μάλλον όλα αυτά τα οποία μας είπε η Κομισιόν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το ημερολόγιο καταστρώματος, ε, για την εμπλοκή των τοπικών ε, κοινωνιών, ε, το γεγονός ότι τα αλλιευτικά θα παρακολουθούνται για τη δραστηριότητά τους σε γενικούς όρους λοιπόν έχουμε μία λογική συμφωνία η οποία λειτουργεί η οποία αποτελεί πρόοδο έναντι των συμφωνιών που ξέραμε μέχρι τώρα και εδώ στο Κοινοβούλιο με τρίτες χώρες. Εμείς πρέπει να αποφασίσουμε τώρα πώς να προχωρήσουμε για το χρονοδιάγραμμα. Εμείς θέλουμε να περιμένουμε μία σταθεροποίηση της κατάστασης στη Γουινέα Μπισάου. Αξίζει τον κόπο διότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια η κατάσταση δεν είναι σταθερή στην ε, Γουινέα Μπισάου και ξέρουμε ότι οι κυβερνήσεις ε, της Γουινέας Μπισάου συνδέονται με, με, με το εμπόριο ναρκωτικών. Δεν είναι καθόλου εύκολη ιστορία δηλαδή η διαπραγμάτευση με αυτές τις κυβερνήσεις. Εμείς θα το κάνουμε βέβαια άμα χρειαστεί δηλαδή να, να έρθουμε πάλι σε επαφές με τις αρχές της Γουινέας Μπισάου σύμφωνοι. Αλλά ας περιμένουμε. να δούμε τι θα γίνει και θα χρησιμοποιήσουμε τον κοινό νου στο τέλος ελπίζοντας ότι το πρωτόκολλο θα μπορέσει να αρχίσει να ισχύει και οι στόλοι μας ε, θα φτάσουν σε αυτά τα χωρικά ύδατα όταν θα το επιτρέπουν οι πολιτικοί και κοινωνικοί όροι. Κυρία Λέβεν. Κυρία πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι πολύ ενισχυτική κατάσταση στην Γουινέα το στρατιωτικό πραξικόπημα και η μεταβατική κυβέρνηση δεν επιτρέπουν ε, την εξέβρεση λύση. Το Συμβούλιο έχει αποφασίσει να μην προχωρήσει διαπραγματεύσεις. Εγώ πρέπει να πω ότι δεν ε, αντιλαμβάνομαι πώς είναι δυνατόν να συνεχίσουμε με την έκθεση αυτή σε τόσο άστατο περιβάλλον. Και όπως είπε και η συγγήτρια, το λαθρεμπόριο των ναρκωτικών στη Γουινέα είναι πάρα πάρα πολύ ανησυχητικό. Έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη χώρα ουσιαστικά και πρέπει να πω ότι για μένα αυτό φαίνεται παράλογο το να μιλούμε για μηνύματα και θεωρήσεις όταν η κυβέρνηση δεν μπορεί τα ύδατά της ε, να ελέγξει. Δεν μπορούν να ελέγξουν τα ύδατα της ε, χώρας η λατινοαμερικανική μαφία των ναρκωτικών έχει ε, απόλυτη κυριαρχία στα εγχώρια τη της χώρας. Και έτσι ενώ μεν είχαμε υπερψηφίσει την προσωρινή ε, παράταση της ισχύου συμφωνίας εν νέων διαπραγματεύσεων, θεωρώντας ότι είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε μια νόμιμη, μια νομιμοποιημένη κυβέρνηση στην Κουίτα Μπισάου, γιατί είναι σημαντική για οικονομικού λόγου για την Κουίνα Μπισάου η συμφωνία αυτή για τον εθνικό του προπολογισμό, υπό τι τρέχουσε συνθήκε και περιστάσει. Θα έλεγα ότι πρέπει μάλλον να περιμένουμε τι εξελίξει να μην προχωρήσουμε. Ευχαριστώ κύριο Σάντες Προσέδου. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες της Κομισιόν. Οι πληροφορίες που είχα εγώ ήταν παλιότερες, από το 80. Η διαπραγμάτευση είχε γίνει πριν από το πραξικόπημα. Και το πραξικόπημα οδήγησε σε ανομαλία και αστάθεια. Το Συμβούλιο διαπραγματε... από με την Αφρικανική Ένωση μετά από συνένεση του ΟΗΕ δεν βλέπω εγώ να μπορέσει ο στόλος μας να συναρχίσει να ψαρεύει στην περιοχή. Και εγώ εκφράζω τη λύπη μου για την κατάσταση. Θεωρώ ότι το πρωτόκολλο θα ήταν ένα καλό πλαίσιο για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας. Αλλά Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παλέψει για, την, για τον εκδημοκρατισμό. Λοιπόν, υπάρχει άλλη τοποθέτηση, κυρία Πατράο. Εγώ δεν ξέρω. Αλλά κυρίως για την τοποθέτηση της κυρίας Λέβιν. Δεν ξέρω αν ήμουν επαρκώς σαφής. Είπα, ας προχωρήσουμε τη δουλειά μας εδώ στο Κοινοβούλιο αναγνωρίζοντας όλα αυτά τα οποία είπε η κυρία Λέβιν, αλλά επειδή πρόκειται για ένα πρωτόκολλο συμφωνίας το οποίο ξεπερνάει τα όρια που το, των πεπραγμένων μας μέχρι σήμερα και έχουμε, έχει ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση Α, εμείς εκφραζόμαστε επ' αυτού το πρωτόκολλου, δεν ξεκινάμε διαπραγματεύσεις ή συζητήσεις με την ε, τωρινή κυβέρνηση που δεν είναι μια νόμιμη κυβέρνηση. Η Πορτογαλία δεδομένου ότι είναι και πρώην ε, απικία μας η Γουινέα Μπισάου, έχει πάρα πολύ σκληρή θέση, δεν αναγνωρίζει καν την κυβέρνηση, αλλά εμείς δεν εκφραζόμαστε εδώ για την κυβέρνηση τη ε, Γουινέας Μπισάου, αλλά για το πρωτόκολλο, το οποίο πρωτόκολλο μαζεύει, ε, συσπηρώνει όλα μας τα ζητούμενα του παρελθόντος, όπου έχουμε και τη ρήτρα για την για την, διασφα... για την ανέρεση του πρωτοκόλου, για παράδειγμα, δεν γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα, λέμε, όπ, ανερούμε το πρωτόκολλο και... και αναστέλουμε λοιπόν την λειτουργία και με την θέση σε ισχύ και μετά το εφαρμόζουμε όταν αλλάζουν τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αποφάσεις των συντονιστών, έχετε τη σχετική, το σχετικό έγγραφο, επόμενη συνεδρίαση 6 Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στις 9. Και ολοκληρώνουμε λοιπόν. Ευχαριστώ όλους σας. Καλό καλοκαίρι. Φορτώστε τις μπαταρίες σας και οι διερμηνείς το ίδιο λέει ο Πρόεδρος. Συμφωνούν οι διερμηνείς. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.